państwa. Wyjaśniłem panu ministrowi. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εξήγησα στον Υπουργό ότι συνήθως ξεκινάμε στις 3 τη συνεδριάσεις μας. Σήμερα λίγο νωρίτερα, στις 2.30. Γι' αυτό και άφησα λίγα λεπτά καθυστέρησης για την έναρξη. Και πριν καλωσορίσω τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, τον Υπουργό Γεωργίας της Ρουμανίας, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι θα ήθελα να εγκρίνουμε πρώτα την ημερήσια διάταξη. Τελικά δεν θα γίνει σήμερα η συνεδρία των συντονιστών, και μία αλλαγή στην ημερήσια διάταξη. Το σημείο 10 που προβλέπει αλλαγή απόψεων με εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα την κατάσταση στην αγορά εσπεριδοειδών θα προηγηθεί του σημείου 9. Δηλαδή τη ανταλλαγή απόψεων με εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το γεωργικό σκέλος των τρεχουσών εμπορικών διαπραγματεύσεων και άλλων θεμάτων της εμπορικής πολιτικής. Υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις για την ημερήσια διάταξη. Ο κύριος Χόισλινγκ. Ο κύριος Χόισλινγκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να διαμαρτυρηθώ γιατί ακυρώθηκε η συνεδρία των συντονιστών. Δεν είχαμε ειδοποιηθεί ε, στην ώρα μας και είχαμε πει ότι σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε να κάνουμε πολλές διαβουλεύσεις γιατί πρέπει να δούμε τη νέα ΚΑΠ. Δεν έχουμε καν ένα χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο, δεν ξέρουμε καν πώς θα ξεκινήσουμε με αυτή την επίγουσα υπόθεση και νομίζω ότι με αυτό το ρυθμό δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Δεν γίνεται. Άρα λοιπόν αναρωτιέμαι, αν θέλουμε να καταλήξουμε σε ένα θεμητό, λογικό αποτέλεσμα. Αν θέλουμε να συνεχίσει να υφίσταται η ΚΑΠ, θέλω να μου πείτε πότε θα ψηφίσουμε και πότε. Και αυτό επρόκειτο να το συζητήσουμε στου συντονιστέ. Με τον τρόπο αυτό που προτείνεται, δεν μπορούμε καν να πούμε ότι εξασφαλίζουμε την αλληλεγγύη. Τα έγγραφα τα λαμβάνουμε λίγη ώρα πριν τη συνεδρίαση. Θέλουμε ένα λογικό ρυθμό εργασία και είναι κάτι το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να συζητήσουμε. Και όχι μόνο αύριο που θα συζητήσουμε με τον Επίτροπο, θα έπρεπε να το έχουμε δει εσωτερικά σε επίπεδο συντονιστών Κύριε Πρόεδρε, εσεί πρέπει να το αποφασίσετε. Θα γίνουν συντονιστέ, δεν θα γίνουν. Γι' αυτό σα ζητώ. Διατηρήστε την ε, συνεδρίαση των συντονιστών έτσι ώστε να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πώ θα ε, προχωρήσουν οι εργασίε μα. Και νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει να το αποφασίσετε εσεί μόνο σα. Θα πρέπει να το αποφύσουμε εμεί εδώ συλλογικά. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε έτσι. Ευχαριστώ κύριος Φλάναγκαν. Συμφωνώ και εγώ με τον προλαλήσαντα. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι αν δεν προβλέψουμε τον κατάλληλο χρόνο για το θέμα αυτό, το αποτέλεσμα δεν θα είναι καλό. Και αν τα επισπεύσουμε και δουλεύουμε άρον-άρον, θα έχουμε συνεδρίαση σχεδόν εισηγητών με τον εισηγητή να μα λέει ότι θα πρέπει πρώτα να το συζητήσω και να συνεννοηθώ με την ομάδα μου και δεν προλαβαίνουν ούτε και εισηγητέ να προετοιμαστεί. Γιατί ακολουθείτε αυτό το ρυθμό και η ιδέα ότι ε, η πλειοψηφία δεν είναι υπέρ τη συνεδρίαση, τότε να μην κάνουμε ποτέ συνεδρίαση των συντονιστών αν αρκεί ένα να αποφασίζει ότι δεν χρειάζεται τέτοια συνεδρία. Έχουμε εκλεγεί, εκπροσωπούμε του ψηφοφόρου μα και δεν μπορούμε ε, κάποια πλειοψηφία να μα μπλοκάρει. Έχουμε ε, αντίστοιχη εμπειρία στη Βόρεια Ελλάδα με τι καθολικέ κοινότητε. Δεν θέλουμε να το βλέπουμε και εδώ. Επειδή είμαστε μειονότητα δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε λόγο. Δικαιούμαστε να έχουμε κι εμεί λόγο. Ευχαριστώ κύριο Σαλμπερντές. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι πολύ συχνό εγώ <laughs> να συμφωνώ με τους προλαλήσαντες, αλλά νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση θα συμφωνήσω και πραγματικά επίγει να κάνουμε μια συνάντηση συντονιστών. Γιατί πρέπει να συζητήσουμε τι πορεία θα ακολουθήσουν οι, εργασίες μας και δεν μου φαίνεται καθόλου σωστό που ακυρώσατε τους συντονιστές. Bardzo dziękuję. Ευχαριστώ. Ε, είχαμε κάνει διαβουλεύσεις με τους συντονιστές και ρώτησα αν χρειάζεται πραγματικά να διατηρηθεί η συνεδρίαση των συντονιστών. Και στις 29 Ιανουαρίου, όπως ξέρετε, θα έχουμε ολοήμερη συνεδρίαση αφιερωμένη στη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Και μετά από γραπτές διαβουλεύσεις που είχα με τους συντονιστές και αφού διαπίστωσα ότι η πλειοψηφία των συντονιστών έκρινε ότι δεν υπάρχει ανάγκη διατήρηση τη συνεδρία, μια και στι 29 Ιανουαρίου θα αφιερώσουμε ολόκληρη τη συνεδρία μα στη μεταρρύθμιση ΚΑΠ, γι' αυτό έλαβε την απόφαση να κυρωθεί η συνεδρία των συντονιστών. και ο ρυθμός που λέτε, το tempo που ακολουθούμε, συνδέεται και παρακολουθεί τις εργασίες για τη μεταρρύθμιση. Δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου που είχαμε για τη μεταρρύθμιση στην αγορά για τα πνευματόδη ή μάλλον συγγνώμη για την βιολογική γεωργία, τότε είχαμε πολύ περισσότερο χρόνο, αλλά πρέπει να προσαρμοστούμε στο χρόνο που έχουμε και να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας, γιατί λόγω της προεκλογικής φάσης αυτής και το ότι τελειώνει η κοινοβουλευτική θετία, είμαστε υποχρεωμένοι να επισπεύσουμε τις εργασίες μας. Η κυρία Σένερα. Ευχαριστώ. Οπότε διαρωτώ με, ποιοι είναι οι συντονιστέ ε, που τάχθηκαν υπέρ τη αναβολή ή τη ακύρωση τη συνεδρίαση. Γιατί εδώ ακούσαμε τρει πολιτικέ ομάδε και οι τρει πολιτικέ ομάδε είναι υπέρ τη συνεδρία των συντονιστών. Εσεί μιλήσετε για γραπτέ διαβουλεύσεις ε, ε, κατά τις οποίες πολλοί συντονιστές αποφάθηκαν κατά τη συνεδρίαση. Ποιοι είναι αυτοί οι συντονιστές που δεν θέλουν τη συνεδρίαση. Έγινε γραπτή διαβούλευση όπως σας είπα. Και από τις ερωτήσεις που έστειλα στους συντονιστές κατέληξα στο συμπέρασμα της απαντήσεως ότι δεν χρειαζόταν ε, να, γίνει, να παραμείνει αυτή η συνεδρίαση των συντονιστών. Από τον αριθμό των απαντήσεων και συγκεντρώνοντας τον αριθμό των ψήφων που εκπροσωπούσαν, έκρινα ότι η πλειοψηφία των συντονιστών δεν ήθελα αυτή την συνεδρίαση. Αλλά τώρα, αν η πλειοψηφία των συντονιστών Ε, είναι υπέρ, ε, το κατανοώ. Ο κύριος Καπούτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ προβληματίζομαι, δεν κατάλαβα. Εγώ απλά έλαβα την ανακοίνωση ότι η συνεδρία των συντονιστών δεν θα λάβει χώρο, δεν χώρα. Όπω είπαν και άλλοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερε συνεδριάσει. Κάπω κάπου υπήρξε κάποια παρανόηση. Εμά μα ανακοινώθηκε ότι δεν υπήρχε τίποτα στην ημερήσια διάταξη και φαινόταν παράλογο να κάνουμε συνέδρια συντονιστών ε, χωρίς ε, ημερήσια διάταξη. Θεωρώ ωστόσο ότι θα πρέπει να το καλύψουμε κάπως αλλιώ, να γίνει κάποια συζήτηση ε, έτσι όπως ήθεστε. Δεν λαμβάνω εγώ την απόφαση για συγκρότηση ή ακύρωση της συνεδρίας των συντονιστών χωρίς τη συμφωνία των συντονιστών. Δεν το, δεν το αποφασίζω μονομερός. Δεν ήταν δική μου απόφαση. Προέκυψε από την πλειοψηφία των ε, συντονιστών. Δεν είναι καμιά δική μου προθυμία ή ε, έλλειψη θέλησης να κάνω τη, συνάντηση. Από τι απαντήσεις των συντονιστών κατέληξα στο συμπέρασμα ότι δεν χρειαζόμασταν αυτή τη συνεδρίαση. Και επαναλαμβάνω, στις 29 Ιανουαρίου θα έχουμε όλη τη μέρα για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Και δεν έχουμε τίποτα ιδιαίτερα μυστικά που θα πρέπει σώνει και καλά να τα συζητήσουμε μόνο μεταξύ μα οι συντονιστέ. Μπορούμε να τα συζητήσουμε ανοιχτά στη δημόσια μα συνεδρία στι 29 Ιανουαρίου. Κύριος Φλάναγκαν. Δεν μ' αρέσει να με θεωρούν λίθιο ρώτησα κάτι και θα ήθελα να απαντήσετε αυτό που σας ρώτησε η συνάδελφος. Ποιοι συντονιστέ σας είπαν πως δεν θέλουν να γίνει η συνάντηση. Δεν μας έχετε δώσει ονόματα. Μέχρι στιγμής ε, το μόνο που έχουμε ακούσει είναι συναδέλφους οι οποίοι παραξενεύονται που ακυρώθηκε συνεδρία. Σας παρακαλώ μην μας περνάτε για ανόητους. Κύριε Ευρωβουλευτά, εγώ δεν είπα ότι κάποιος συγκεκριμένος συντονιστής ζήτησε να ακυρωθεί η συνεδρίαση των συντονιστών. Απλώς εγώ ρώτησα, υπάρχει λόγος να γίνει συνεδρίαση. Και δεν υπήρχε πλειοψηφία υπέρ της διοργάνωσης της συνεδρίασης. Γι' αυτό και αποφάσισα να την αναβάλω. Εγώ ρώτησα και κανένας συντονιστής δεν επέμεινε να γίνει. Απλώς ρώτησα. Από τη στιγμή που δεν έχουμε θέμα, υπάρχει λόγος να γίνει συνεδρίαση. Και επειδή δεν βρέθηκε πλειοψηφία να ζητά τη συνεδρίαση, γι' αυτό αποφάσισα να την αναβάλω. Δεν είναι ότι εγώ δεν ήθελα να συζητήσουμε συντονιστέ. Αλλά μια και δεν έλαβα απάντηση όταν ρώτησα υπάρχουν θέματα προς συζήτηση, θεώρησα ότι η σιωπή δηλώνει ότι δεν υπάρχουν αρκετά θέματα. Από τη στιγμή που δεν μπήκατε στον κόπο να απαντήσετε στι ερωτήσει μου, σημαίνει ότι δεν ε, υπήρχε λόγος για τη συνεδρίαση. Κύριε κύριος Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη, ε, καθυστέρησα λίγο, αλλά ακούσαμε τώρα ο συντονιστή του ΕΛΚΕ είπε να λάβει ο Σοσιαλιστή επίση, ο συντονιστή των Πρασίνων επίση και τη Γκουε, όλοι αυτοί ζητάνε να λάβει χωρέ συνεδρίαση. Υπάρχει πλειοψηφία και εμένα μου κάνει έκπληξη διότι τελικά ε, πλησιάζουμε στο τέλο τη θετίας και ξαφνικά ακυρώνουμε ενώ υπάρχει ένα ε, αίτημα από την πλειοψηφία να γίνει συνεδρίαση. Δεν καταλαβαίνω πού μπλόκαρε η κατάσταση, για ποιο λόγο. Και εγώ υπήρξα συντονιστή στο παρελθόν. Γιατί να μην λάβει χώρα αύριο, όπω γίνεται. Τελικά δεν είναι δική μου υπόθεση, είναι, ε, από εσά εξαρτάται, αλλά αν υπάρχει βούληση να λάβει χώρα η συνεδρία, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο ότι σταματάει κάποιο. Ε, κάποια λίγο βούληση χρειάζεται να ολοκληρώσουμε αυτή τη θητεία ε, κανονικά και ήρεμα. Ε, πώς, Κύριε Ευρωβουλευτά, αξιότιμοι συνάδελφοι, τη διαβούλευση την έκανε η γραμματεία εκ μέρους μου. Οπότε θα ζητήσω από το Γενικό μας Γραμματέα να απαντήσει. Γιατί δεν έκανα εγώ προσωπικά τις ερωτήσεις του συντονιστές. Κυρία Μίλλερ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας πω πως καταλαβαίνω το εξής. Πραγματικά τα συναισθήματα είναι έντονα, αλλά εγώ όντως το φθινόπωρο είπα πως χρειαζόμαστε ένα χρονοδιάγραμμα για την ΚΑΠ, για να είναι τα πράγματα ξεκάθαρα. Και δεν υπερψηφίστηκε. Και τελικά τι γίνεται, καθυστερούμε, μεταφέρεται από τη μία συνεδρίαση στην άλλη. Νομίζω πως την Τρίτη θα πρέπει να συναντηθούν οι συντονιστέ. Και εκεί, μαζί με τους συντονιστές, να δούμε και τους τρεις εισηγητές για να εξετάσουμε το θέμα, για να ψηφίσουμε. Επιτέλους, έχω τέσσερις μήνες που περιμένω να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Φτάνει πια. Λοιπόν, για του υπόλοιπου συντονιστέ, να σας πω ένα καλό νέο. Εγώ πια δεν είμαι συντονιστή, γιατί άλλαξα ομάδα πολιτική στο Στρασβούργο την, την προηγούμενη φορά. Οπότε ίσως αυτό να σας βοηθήσει. Αλλά νομίζω ότι τελικά σε αποτέλεσμα με αυτό το ρυθμό δεν θα φτάσετε. E, Ευχαριστούμε γιατί συμβάλλετε να δημιουργηθεί μια πιο ελαφριά ατμόσφαιρα, ένα κλίμα πιο θετικό. Ναι, ακούστε, η κατάσταση είναι λίγο λεπτή. Κάπου υπήρξε κάποια παρανόηση, φαντάζομαι. Εγώ πολύ ειλικρινά και με διαφάνεια θα σας διηγηθώ τι συνέβη για αυτή τη συνεδρία των συντονιστών. Ουσιαστικά η διαδικασία υπήρξε η συνήθις. Ε, αναφέρουμε στη γραμματεία ένα κατάλογο με τα θέματα για τα οποία θα κληθούν οι συμμετέχοντες να λάβουν αποφάσεις, ε, αποφάσεις εκθέσεις, ε, και παρουσιάσαμε αυτό τον κατάλογο με τους συναδέλφους και είδαμε ότι ελάχιστα ήταν τα θέματα. Υπήρχε μία μόνο ουσιαστικά απόφαση, η έγκριση του χρονοδιαγράμματος των τακτικών συνεδριάσεων της Επιτροπής Γεωργίας για το δεύτερο μισό του έτους. Μία απόφαση που μπορεί να ληφθεί πανεύκολα με τη γραπτή διαδικασία. Υποβάλαμε λοιπόν ε, στον πρόεδρο ε, αυτή την, αυτά τα σημεία, αυτό το κατάλογο, λέγοντα ότι δεν υπάρχουν αρκετά σημεία, βλέποντα αν θα πρέπει να γίνει συνεδρίαση ή όχι. Και τελικά έγινε διαβούλευση με του συντονιστέ, όλοι λάβατε ένα μήνυμα όπου σα εξηγούσαν ότι ήταν ελάχιστε οι αποφάσει και προτινόταν ενδεχομένω να ακυρωθεί η συνεδρίαση και από αυτή τη διαβούλευση λάβαμε μόνο τρει απαντήσει, αν δεν κάνω λάθο. Μία από την ομάδα των Πρασίνων πράγματι που ζητούσε να γίνει η συνεδρίαση ούτως ή μια απάντηση από την ΚΟΕ που... και μετά μια απάντηση από την ομάδα του ΕΛΚΑ. Οι άλλες ομάδες στη συνέχεια, από όσο ξέρω, δεν απάντησαν σε αυτή τη διαβούλευση. Αυτά τα παρουσιάσαμε εμείς στον πρόεδρο, βάσει των οποίων ελήφθη η απόφαση να ακυρωθεί η συνεδρίαση των συντονιστών. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο έπαιξε ρόλο για να διορθώσω αυτά που υπόθηκαν ότι την Τρίτη το απόγευμα, την περασμένη εβδομάδα, στις... Ε, ζητήθηκε ε, η συνεδρίαση της ε, Επιτροπής Γεωργίας να αφιερωθεί αποκλειστικά στην ΚΑΠΑ, να δούμε τις τροπολογίες, τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠΑ, και αυτό έπαιξε ρόλο στο να αποφασίσουμε να πούμε ότι τελικά δεν ήταν τόσο αναγκαίο να γίνει ε, η συζήτηση αυτή τη συνέδρια των συντονιστών, αλλά όπως είπα είχε προβλεφθεί μια ανοιχτή ε, συνεδρίαση της Επιτροπής Γεωργίας και όχι συνεδρίαση συντονιστών. Αυτά συνέβησαν, σε αυτό το στάδιο βρισκόμαστε. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Ε, ε, μια στιγμή μετά από δική μου παράκληση, ρητή παράκληση, έγινε γραπτή διαβούλευση για να μην με κατηγορήσουν οι συντονιστέ ότι έλαβα μονομερό την απόφαση. Μετά από δική μου παράκληση, η γραμματεία έκανε γραπτή διαβούλευση με τις ομάδες. Οπότε με κατηγορείτε ότι δεν ήθελα να γίνει συνεδρίαση. ότι δεν ήθελα να κάθομαι εδώ συνεδρίες των συντονιστών ή γιατί δεν είχα χρόνο ή δεν είχα διάθεση να διοργανώσω την συνεδρία στο Συντονιστό. Ο κύριος Χόισλινγκ. Εμείς θα θέλαμε να ακούσουμε εδώ και τον κύριο Υπουργό. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την ε, συζήτηση, την ατέρμονη, οπότε ή αν πρόκειται για παρανόηση, εντάξει. Αυτό το οποίο όμως δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να ψηφίσουμε ε, το χρονοδιάγραμμα σε αυτή τη δημόσια συζήτηση που θα κάνουμε την επόμενη εβδομάδα. Θα πρέπει αυτό να γίνει στους συντονιστές ε, με τους εισηγητές. Άρα λοιπόν θα στηρίξω την κυρία Μίλλερ την επόμενη εβδομάδα να συνεδριθούν οι συντονιστέ, γιατί εκεί πρέπει να λύσουμε το θέμα του χρονοδιαγράμματο. Ε, και νομίζω είναι κάτι το οποίο θα χρειαστεί πάνω από πέντε λεπτά. Γιατί, επαναλαμβάνω, πρέπει τα πράγματα να είναι σαφή, να είναι καθαρά. Οπότε, εντάξει, σήμερα όχι, αλλά την επόμενη εβδομάδα ναι. Και όταν λέω δεν μπορούμε να το συζητήσουμε το θέμα αυτό στην ανοιχτή συζήτηση, Το λέω γιατί είναι εσωτερικό πρόγραμμα εργασιών με τους τρεις συγητές. Μάλιστα. Πάντως ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να διοργανώσουμε τελικά τη συνεδρία των συντονιστών ε, παρόλο που δεν είχαμε προγραμματίσει, να έχουμε χρόνο και διερμηνία. Και πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να επανερχόμαστε συνέχεια στη συζήτηση για τις υποχρεώσεις μας. Το συζητήσαμε το θέμα, βγήκε ένα χρονοδιάγραμμα, διαπιστώσαμε ότι χρειάζεται μια επίσπευση των εργασιών, είναι φορτωμένο το πρόγραμμα και αυτό μπορεί να επιβαρύνει λίγο τους συγητές και τους κοιόδης συγητές, αλλά αυτό έχει αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν έχει νόημα τώρα να το συζητάμε. Θα περάσουμε στην ακρόαση με τον Υπουργό Γεωργίας της Ρουμανίας, στην ανταλλαγή απόψεων. Δεν ήταν και μυστικό ε, αυτό που ακούστηκε στη συζήτηση και στη, στο Συμβούλιο Γεωργίας θα έχει αρκετά δύσκολε συζητήσει ο Υπουργό. Ξέχασα να σα πω ότι έχουμε και διερμηνία σε 20 γλώσσε και ότι μεταδίδεται από το διαδίκτυο η συνεδρίασή μα. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Υπουργό που είναι πολύπειρος γιατί και στο παρελθόν διατέλεσε Υπουργό Γεωργίας το 2004, ήταν και Υφυπουργό, είχε διάφορες ιδιότητες και είχε αναλάβει διάφορα καθήκοντα ε, και θα αντιμετωπίσει τώρα προκλήσει στα πλαίσια τη Προεδρία. Μάλιστα, το σύνθημα τη Ρουμανική Προεδρία είναι η συνοχή, μια κοινή ευρωπαϊκή αξία. Κάτι που ε, αντανακλά την ιδέα μια Ευρώπη ενότητα και ε, αλληλεγγύη που εκτιμούμε ιδιαίτερω. Οπότε, στα πλαίσια τη Ρουμανική Προεδρία θα συζητήσουμε για την ΚΑΠ μετά το 2020, για τι δημοσιονομικέ προοπτικέ, το νέο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και μια σειρά προβλημάτων. Γιατί όπως ξέρετε έχουμε πάρα πολλές ε, τροπολογίες. Έχουμε καταρχήν την έκθεση για τα εθνικά στρατηγικά σχέδια. Πολλοί άνθρωποι είναι τροπολογίε που έχουν κατεθεί, κατατεθεί και εκεί. Φαντάζομαι θα τα σχολιάσετε όλα αυτά στην ομιλία σα. Σα καλωσορίζω εγκαρδιότατα και θα ήθελα να σα δώσω το λόγο. Και σα δώσω συγγνώμη που χρειάστηκε για να γίνετε μάρτυρα σε αυτών των εσωτερικών μα ε, συζητήσεων. Ε, και καθυστερήσαμε και όλα τη δική σας συζήτηση. Χρειάστηκε να τα ακούσετε και αυτά. Εν πάση περιπτώσει, αυτά έχει ζωή. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ δεν έχω δώσει ε, τίποτα σε αυτή τη συζήτηση ως συνεισφορά, αλλά η δική μου ε, εμπειρία μου ε, έχει επιτρέψει να λάβω, χώρα, να λάβω μέρος στη συνεδρίαση σήμερα να δω τι θα μπορούσα και εγώ να σας πω. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ Άνταμ, κύριοι ευρωβουλευτές, κυρίες ευρωβουλευτές. Είναι για μένα πραγματική τιμή και χαρά να είμαι εδώ σήμερα μπροστά σας για να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Ρουμανικής Προεδρίας ε, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να ξεκινήσω μεταφέροντας τα, ε, τους χαιρετισμού των γεωργών από τη Ρουμανία που έχουν ευνοηθεί από την ΚΑΠ και εσείς έχετε συνεισφέρει στην πολιτική αυτή και ξέρω πώς θα το κάνετε ε, και στα πλαίσια της ε, κοινή πολιτικής για την περίοδο 21-27 γιατί η Ρουμανία είναι, είναι μια στιγμή πάρα πολύ σημαντική είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνουμε ε, προεδρία και είναι 12 χρόνια μετά τη στιγμή της ένταξής μας. Πες περιμένει λοιπόν μια περίοδος πολύ δυναμική με σημαντικές εκδηλώσεις για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι εκδηλώσεις οι οποίες σύντομα έρχονται και θα ήθελα να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να ε, εκπληρώσουμε ε, τη ρόλο μας που είναι ε, το να είμαστε ένας αντικειμενικός επιδιαιτητής που θα μας ε, βοηθήσει να προχωρήσουμε στην οικοδόμηση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Έχουμε τη διάσκεψη της, ε, του CBU το Μάιο που θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε σε μια πιο δημοκρατική Ευρώπη με περισσότερη συνοχή. Είναι μια συνάντηση σε υψηλό επίπεδο που θα επιτρέψει να ευαισθητοποιήσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες για τα απτά αποτελέσματα των αποφάσεων που λαμβάνονται στο επίπεδο της αλλά και για τι απαραίτητε μεταρρυθμίσει για να συνεχίσουμε να προοδεύουμε και να ενισχύουμε και να ενδυναμώνουμε το ευρωπαϊκό σχέδιο. Θέλουμε η δική μας Προεδρία να ε, στραφεί προς τους πολίτες και για το λόγο αυτό θα ήθελα, ε, θα θέλαμε να ε, τους επικοινωνήσουμε το ευρωπαϊκό θεματολόγιο και να καταλάβουν γιατί τους αφορά. Μέσω ε, της δράσης που θα έχουμε ως Προεδρία του Συμβουλίου θέλουμε να πετύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα και να ε, υπογραμμίσουμε τα πλεονεκτήματα που προσφέρει μια δυνατή ένωση με περισσότερη συνοχή σε όλους μας. Παράλληλα η Προεδρία θα έχει πάντα υπόψη της το ότι η ευρωπαϊκή πολιτική θα πρέπει να ακολουθεί την αρχή της ε, ε, ισότητας και της συνοχής μεταξύ περιοχών, περιφερειών και πολιτών. Η συνοχή είναι στο κέντρο της ε, πολιτικής μας και είναι η κοινή ευρωπαϊκή μας αξία. Οι προτεραιότητες μας είναι τα εξή. Η Ευρώπη της σύγκλησης, η Ευρώπη της ασφάλειας, η Ευρώπη ε, παγκόσμιος παίκτη και η Ευρώπη και οι κοινέ μα αρχέ. Για τον πρώτο από αυτού του πυλώνες θα ήθελα να σα πω πω ο βασικό μα στόχο είναι η σύγκληση και η συνοχή στην Ευρώπη, έτσι ώστε να είναι βιώσιμη ανάπτυξη, να είναι δίκαιη ανάπτυξη για όλου τους πολίτες και για όλα τα κράτη-μέλη, αυξάνοντα την ανταγωνιστικότητα και μειώνοντα τι διαφορέ που έχουμε στα αναπτυξιακά επίπεδα, στην κοινωνική πρόοδο, με καλύτερη διασυνδεσιμότητα, με ψηφιοποίηση και προωθώντα το επιχειρήν όπως επίσης και τη βιομηχανική πολιτική. Δεύτερος πυλώνας. Η βασική αρχή είναι η Ευρώπη της ασφάλειας. Και για να παγιωθεί η ασφαλής Ευρώπη με μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των κρατών μελών, μια και αντιμετωπίζουμε νέες προκλήσεις στην ασφάλεια και νέες απειλές προς τους πολίτες μας, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε πρωτοβουλίες συνεργασίας, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Τρίτος πυλώνας. Εκεί ο βασικός μας στόχος είναι η Ευρώπη να γίνει ένας παγκόσμιος παίκτη. Να ενισχυθεί ο ρόλος μας στην παγκόσμια σκηνή και να εφαρμόσουμε την ε, παγκόσμια μας στρατηγική έτσι ώστε να έχουμε τους απαραίτητους πόρους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και προωθώντας την πολιτική της διεύρυνσης όπως επίσης και της ε, γειτονίας έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στους, ε, στις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μιλήσω τώρα για τον τέταρτο πυλώνα όπου γενικότερο στόχος μας είναι να προκρίνουμε και να προωθήσουμε την αλληλεγγύη και τη συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι θα προωθήσουμε τη μάχη για να καταπολεμήσουμε την ανισότητα, την, ε, τις άνισες ευκαιρίες, θα προωθήσουμε την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και θα ανοίξουμε την ευρωπαϊκή συζήτηση στους Ευρωπαίους πολίτες. Η δική μας Προεδρία θα περιγράψει τις αρχές του επόμενου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027. Αυτός ο μελλοντικό προϋπολογισμός θα πρέπει να προσφέρει τους απαραίτητους πόρους για να πετύχουμε τους στόχους μας για τα επόμενα 7 έτη έχουμε δεσμευθεί σε επίπεδο προεδρίας και σε πολιτικό επίπεδο και σε τεχνικό επίπεδο να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα στο Συμβούλιο και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε να πετύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα κλείνοντας αυτές τις διαπραγματεύσεις με μεγαλύτερη σύγκληση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο στόχος αυτός είναι μια προτεραιότητα για μας και στιγμή αφετηρίας για όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πολιτικές. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά τη σημασία που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια και εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους πολίτες και λαμβάνοντας υπόψη τη μακρά μου κοινοβουλευτική εμπειρία, σε, πήρα με συγχωρείτε, σε εθνικό επίπεδο, γιατί ήμουνα και στην δική μας, στο δικό μας κοινοβούλιο μέλος της Επιτροπής Γεωργίας και πρόεδρος αυτής για τέσσερα χρόνια. Για το λόγο αυτό μπορώ να σας επιβεβαιώσω πως έχω κάθε διάθεση να συνεργαστώ μαζί σας με επικοδομητικό τρόπο, με αποτελεσματικό τρόπο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε ε, αυτή την πορεία προόδου όπως έχει γίνει και με τις προηγούμενες προεδρίες. Η ομάδα μου και εγώ είμαστε στη διάθεσή σας και στο πνεύμα της συνεργασίας δεσμευόμαστε να δουλέψουμε μαζί σας. Μια και είμαι εδώ λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Κέστιγκερ και την ομάδα της για όλες τις ε, προσπάθειες που έκανε και τις επιτυχίες που σημείωσε μέχρι σήμερα. Θα ήθελα επίσης Άνταμ και σένα να σε συγχαρώ και σένα και την ομάδα σου για το ρεαλιστικό και αποτελεσματικό τρόπο με τον οποίο έχεις ε, διευθύνει τις διαπραγματεύσεις μέχρι σήμερα. Έχω την ελπίδα πως θα συνεχίσουμε έτσι για όλους τους φακέλους που είναι αυτή τη στιγμή σε εκκρεμότητα. Θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Να δούμε την πραγματικότητα κατάματα, γιατί έχουμε πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία και για να κλείσουμε με όλες τις διαδικασίες έγκρισης των νομοθετικών σχεδίων πριν τις ευρωεκλογέ. Ξέρετε πως ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός και είναι μια τεράστια πρόκληση για όλους τους θεσμούς, αλλά είμαι σίγουρος πως θα πετύχουμε. Αυτή τη στιγμή ε, έχω να σας πω πως οι υπηρεσίες του Συμβουλίου έχουν οργανώσει σωστά τη δουλειά τους και για το νομοθετικό πακέτο για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ μέσα στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο είναι η βασική προτεραιότητα της δικής μας προεδρίας. Τουλάχιστον για τα όσα θα συμβούν στον κλάδο της γεωργίας. Θέλουμε λοιπόν να συνεχίσουν οι συζητήσεις για το πώς μπορούμε να εξυγχρονίσουμε και να απλουστεύσουμε την ΚΑΠ, λαμβάνοντας υπόψη πώς η διαδικασία αυτή θα πρέπει να σεβαστεί πλήρως όλες τις διατάξεις που έχει η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τον ουσιαστικό ρόλο που έχει η κοινή αγροτική πολιτική για να γίνει πιο ανταγωνιστική η Ευρωπαϊκή Ένωση και πόσο απαραίτητη είναι ο χρονισμός και η απλούστευση. Αυτά μπορούν ε, να οδηγήσουν σε μια πιο αποτελεσματική ΚΑΠ που θα εξασφαλίσουν ένα επίπεδο ζωής που θα είναι δίκαιο για τους γεωργικούς πληθυσμούς στην Ήπεθρο με εξασφαλισμένη διατροφική ασφάλεια, με λογικές τιμέ για τα τρόφιμα για όλους, αυξάνοντα δε την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τον ειδικό, τον ιδιάζοντα χαρακτήρα της ε, γεωργίας σε κάθε κράτος που βασίζεται στις κοινωνικές δομές κάθε κράτους όπως επίσης τις ε, φυσικές ή διαστροτικές ε, διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Εάν θέλουμε ο στόχος μας να είναι μια κοινή αγροτική πολιτική που θα είναι πιο καλά προσαρμοσμένη στις προκλήσεις του μέλλοντος Εάν θέλουμε να έχουμε μια πολιτική που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις απαιτήσει όλων των κρατών μελών, τότε θα πρέπει να συνεχίσουμε με τη διαδικασία της νομιθετικής προετοιμασίας. Και αυτό αποτελεί στόχο βασικό της Προεδρίας μας λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη και σε απόλυτο συσχετισμό τότε ότι τρέχουν αυτή τη στιγμή διαπραγματεύσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο ε, για την περιοδο 2021 21-27. Η Ρουμανική Προεδρία θα συνεχίσει να συμμετέχει και να προωθεί τη συζήτηση έτσι ώστε να έχουμε συνένεση για τα κοινά σημεία ε, της αρχιτεκτονικής της, ε, της ΚΑΠ του μέλλοντος. Θέλουμε να έχουμε μια γενική προσέγγιση, μερική έστω, για τα όσα θα γίνουν με το πακέτο αυτό. Και γι' αυτό θα οργανώσουμε συζητήσεις έτσι ώστε να συνεχίσουμε τις προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και για να εντοπίσουμε νέες λύσεις έτσι ώστε τα, πρωτεϊνούχα η, τα πρωτεϊνούχα φυτά, για παράδειγμα, και η καλλιέργεια αυτών να προωθηθεί και ε, να έχουμε φυτικές πρωτεΐνες επαρκής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, εξωτερική σύγκληση για τις άμεσες ενισχύσεις, απλούστευση και περισσότερη επικουρικότητα στα κάτι μελη Έτσι ώστε να έχουμε αυτές τις, ε, ε, ε, αυτά τα σχέδια ανάπτυξης που θα προσαρμόζονται καλύτερα στις ιδιάζουσες συνθήκες τους. Για μένα, οποιαδήποτε στρατηγική για το μέλλον ε, της γεωργίας θα πρέπει επίσης να λάβει υπόψη την ηλικιακή ανανέωση και το ότι η μία γενιά διαδέχεται την άλλη. Για να βρουν μια γεωργία την οποία εμεί χειριζόμαστε καλύτερα, έτσι ώστε να μπουν και καινούριε γενιέ στη γεωργία και για να μην ε, εγκαταλείπονται πλέον οι ζώνε τη υπαίθρου από του νέου και να μην έχουμε αυτή την γύρανση του γεωργικού πληθυσμού, που είναι μια διαδικασία ε, πολύ επικίνδυνη ε, για τη γεωργία. Παράλληλα, θα πρέπει να στηρίξουμε τους μικρούς γεωργούς, τους μικρούς παραγωγούς, οι οποίοι διατηρούν εν ζωή αυτές τις ζώνες ε, ε, της Υπέτρου και κυρίως τις ορεινές, όπου έχουμε πολλούς νέους γεωργούς. Αυτοί θα ε, επιτρέψουν να έχουμε μεγαλύτερη σύγκληση στις ζώνες αυτές στην Ευρώπη, έτσι ώστε να κάνουν έρευνα, να αναπτύξουν νέα προϊόντα, να δούμε τη βιολογική καλλιέργεια. Όλα αυτά θα συζητηθούν και σε επίπεδο Συμβουλίου το πρώτο τρίμηνο. Γιατί αν δεν έχουμε έρευνα, αν δεν έχουμε ε, ε καινούργια στοιχεία, δεν θα καταφέρουμε να βρούμε ε, πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε ε, καλύτερα τους στόχους μας. Η βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Γεωργία. Η διαφύλαξη της ικανότητάς μας να ανταποκρινόμαστε σε όλο και πιο περίπλοκες προκλήσεις απαιτεί ισότιμη πρόσβαση στη χρηματοδότηση για την έρευνα για όλα τα κράτη-μέλη, όπου και αν βρίσκονται γεωγραφικά. Και σίγουρα η βιοοικονομία θα παίξει κέριο ρόλο σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τις συνέργειες μεταξύ των διαφόρων πολιτικών. Θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τα αποτελέσματα της έρευνας και να ενθαρρύνουμε την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών και ιδεών προκειμένου να μειώσουμε τις απώλειες και τη σπατάλη των τροφίμων και ταυτόχρονα διαφυλάξουμε τους φυσικούς μας πόρους. Όλα αυτά φυσικά θα απαιτήσουν Ε, την, ε, τους κανονισμούς 1305-1306 του 2013 για τη χρηματοδότηση ε, και την ΚΑΠ 1307 του 2018 για τις, ε, για τις άμεσες ενισχύσεις και την 1308 του 2013 για την κοινή οργάνωση αγορών. Όλοι αυτοί οι κανονισμοί 1305, 06, 07 και 08 του 2013 θα πρέπει να τροποποιηθούν σε ό,τι αφορά τους κανονισμούς 1305 και 1307 ε, του 2013 για τις άμεσες ενισχύσεις και την ε, ε, στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 2019 και 2020. Αυτός ο κανονισμός έχει, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση των μέτρων στους πυλώνες 1 και 2 για την διετία που σας ανέφερα, το 2019 και το 2020. Θα πρέπει μεταξύ άλλων να επιτρέψει τα κράτη-μέλη να μεταφέρουν κονδύλια μεταξύ των δύο πυλώνων και το 2020 και να ισχύσουν πιο γενναιόδορες ε, συνθήκες ε, και προϋποθέσεις ειδικά για τις ζώνες με φυσικούς περιορισμούς. Και θα μπορεί να γίνει χρήση των κονδυλίων τεχνική τεχνικής αρρωγής για την κατάρτιση των στρατηγικών σχεδίων. Εδώ η Ρουμανική Γεωργία έχει λάβει την ομόφωνη υποστήριξη των κρατών μελών στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας του Συμβουλίου και μάλιστα έχει στείλει επιστολή σύμφωνίας ε, προς τον Πρόεδρο Σεκέρσκι της Επιτροπής σας. Ελπίζουμε λοιπόν η διαδικασία αυτή να διεκπαιρεωθεί αισίω το συντομότερο δυνατό. Η οδηγία για την καταπολέμηση των αθέμητων εμπορικών πρακτικών είναι ένα άλλο σημαντικό θέμα. Έγιναν οι διαπραγματεύσει στα πλαίσια του τριμερού διαλόγου μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων και, στις, και στις, ε, το Δεκέμβριο του 2018 καταλήξαμε σε συμφωνία. Και χαίρομαι γι' αυτό. Η Ρουμανική Προεδρία θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προετοιμάσει την οριστική συμφωνία ώστε η οδηγία για την πάταξη των αθέμητων εμπορικών πρακτικών να ε, τεθεί σε ισχύ πριν το πέρα τη κοινοβουλευτική σα θητεία. Και προσβλέπω εδώ στη συνεργασία, στη στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί η οδηγία αυτή είναι πολύ σημαντική. Και η Ρουμανική Προεδρία, όπως σα είπα, έχει ήδη εξασφαλίσει τη συμφωνία της Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας, όπως έχει επιβεβαιωθεί στην επίσημη επιστολή που εστάλει στον πρόεδρό σας, τον κύριο Σεκέρσκι. Και ευελπιστώ ότι η διαδικασία αυτή θα διεκπαιρεωθεί και επισήμως το συντομότερο δυνατόν. Γνωρίζω το θέμα τη οδηγία για την καταπολέμηση των αθέμητων εμπορικών πρακτικών, τα προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα κάνουμε πραγματικά τη διαφορά στην αγορά και για του γεωργού, αλλά και για του άλλου κρίκου τη αλυσίδα ε, εφοδιασμού σε τρόφιμα και έχουμε πια ένα εύρυθμο εργαλείο για να καταπολεμήσουμε τις μονομερείς καταχρήσεις εκ μέρους κάποιων διανομέων και θέλουμε μία αλυσίδα παροχής τροφίμων ε, που θα διέπεται από αρχές και κανόνες και θα είναι ίσο δίκαιη και για τους γεωργούς. Ένα άλλο σημαντικό νομοθετικό ζήτημα αφορά τα ενοπνευματόδη ποτά και τη ρύθμιση για τα ενοπνευματώδη η Ρουμανική Προεδρία θα πράξει τα δέοντα ώστε ο σχετικό κανονισμό να εγκριθεί πριν το πέρα τη κοινοβουλευτική αστητεία. Και εδώ φυσικά υπολογίζω στη δική σα συνεργασία για να ολοκληρώσουμε τι απαραίτητε διαδικασίε και να τεθεί σε ισχύ ο σημαντικό αυτό κανονισμό για τα εινοπνευματόδη. Σα διαβεβαιώ ότι είμαστε πρόθυμοι για συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα ήθελα και οι μεταποιητές ε, τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης να απολαμβάνουν μια κοινή γεωρική πολιτική που θα ανταπεξέρχεται στην αποστολή της και θα πληρεί τους στόχους της. Το θέμα της καλής μεταχείρισης των ζώων είναι επίσης μείζον μέλημα και της κτηνοτροφίας ε, και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι που είναι και ζωτική σημασία για την οικονομική ανάπτυξη των κρατών μελών και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ρουμανική Προεδρία θα συνεχίσει τι συζητήσει για σημαντικέ επιδημίες και ζωονόσους που μετατρέπονται, που μεταδίδονται διασυνοριακά. Και σίγουρα η Αφρικανική Πανόλη το χείρο ήταν μια τέτοια ε, επιζωτία που μας προβλημάτισε το περασμένο χρόνο. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις οικονομικές συνέπειες που προκάλεσε η επιζωτία αυτή στην ε, Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Και η Ρουμανική Προεδρία θα διευκολύνει τις συζητήσεις για την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων στο Συμβούλιο και στην Υπουργική Διάσκεψη που θα λάβει χώρα στο Βουκουρέστι με το θέμα αυτό, αλλά και το θέμα των ε, άλλων ζωονόσων που μεταδίδονται διασυνοριακά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε τεχνικό επίπεδο, η Ρουμανική Προεδρία θα προωθήσει τη συζήτηση για μια ομοιόμορφη προσέγγιση για να εμπεδώσουμε τις ικανότητες πρόληψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, και μάλιστα να εφαρμόζονται με ομοιόμορφο τρόπο σε όλα τα κρατη Θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην βιοασφάλεια γενικώ, γιατί χάρη στη βιοασφάλεια θα μπορέσουμε να προλάβουμε ασθένειες και να προστατεύσουμε και την υγεία των ζώων. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η μικροβιακή αντοχή και η στρατηγική μας για τη μικροβιακή αντοχή. Η Ρουμανική Προεδρία θα προωθήσει την ε, προσέγγιση της ενιαίας υγείας, One Health. Και μάλιστα θα πρέπει να προσδιορίσουμε τη μελλοντική μας πορεία, τα μελλοντικά μας βήματα Γι' αυτό και θα οργανώσουμε σχετική υπουργική διάσκεψη στο Βουκουρέστι για το θέμα της μικροβιακής αντοχής. Η ευζοία, η καλή μεταχείριση των ζώων, επαναλαμβάνω, είναι σημαντικό θέμα για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα εξετάσουμε τις συστάσεις του ελεκτικού συνεδρίου για την καλή μεταχείριση των ζώων, για να καλύψουμε το κενό μεταξύ των φιλόδοξων στόχων μας και της ε, ανεπαρκούς εφαρμογής και θα προωθήσουμε τις, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για το θέμα αυτό. Επίση, εξαγωγή ζώων των ζώων θα εξακολουθεί να είναι σημαντικό, σημαντική πηγή εισοδήματο για του ε, Ευρωπαίου κτηνοτρόφου. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τη συζήτηση για να εντοπίσουμε τι καλέ πρακτικέ και να προωθήσουμε λύσει για να εξασφαλίσουμε καλή μεταχείριση των ζώων και κατά τη θαλάσσια μεταφορά του. Και ένα σχετικό σεμινάριο μάλιστα θα διοργανωθεί στο Βουκουρέστι παράλληλα με μια άτυπη συνεδρίαση των επικεφαλής κτηνιατρικών υπηρεσιών που θα γίνει τον Ιούνιο. Η διαχείριση των ε, δασών είναι ένα άλλο σημαντικό θέμα για τη Ρουμανία. Η προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές απαιτεί μια ε, αηφόρο βιώσιμη διαχείριση των δασών. Κάτι που αποτέλεσε σημαντικό θέμα προσυζήτηση στην Ευρώπη και διεθνώς. Η Ρουμανία έχει μακροχρόνια πείρα και τεχνικές γνώσεις για τη βιώσιμη διαχείριση των δασών. Η προσέγγιση μας λοιπόν θα στηριχθεί στην προσπάθεια της προσαρμογής του δασικού κλάδου στις κλιματικές αλλαγές, στις κοινωνικές αλλαγές, προκειμένου να αποφύγουμε την υποβάθμιση του εδάφους. Και υπάρχουν πολλές πολιτικές και τομεακά εργαλεία και μέσα που ε, επηρεάζουν τη δασική πολιτική δεν υπάρχει μια αμυγή δασική πολιτική. Αλλά να λιάνεται και με τις άλλε. Εμείς πιστεύουμε ότι η δασική πολιτική θα πρέπει να ρυθμίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με μια διατομεακή προσέγγιση. Η ισχύουσα στρατηγική ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ε, βιώσιμη διαχείριση των δασών 2018-2020 αλλά και η πολιτική μετά το 2020 θα πρέπει να εξασφαλίσει συνέργεια μεταξύ των διαφόρων κλάδων και να συμπεριλαμβάνει ε, σε κοινή συζήτηση τις ε, τομεακές πολιτικές που επηρεάζουν τη διαχείριση των δασών. Μία νομικά δεσμευτική συμφωνία για τα δάση θα συμβάλλει κατά τη γνώμη μας ε, στην υλοποίηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης για το 2030. Οι προηγούμενες προεδρίες, η Βουλγαρική και η Αυστριακή, εργάστηκαν σκληρά προκειμένου να σημειώσουμε πρόοδο στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Δάση. Εμεί θα προωθήσουμε περαιτέρω αυτή τη στρατηγική, προκειμένου να, να καταλήξουμε σε κοινέ προδιαγραφές για βιώσιμη διαχείριση των δασών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο ισχύον διεθνέ πλαίσιο απαιτείται ομοφωνία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ε, αποφαθούμε με ενιαία φωνή στο 14ο Διεθνές Φόρουμ για τα δάση που θα λάβει η χώρα ε, φέτος. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και ενιαία φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ για την ε, πολύπρευρη παρουσίαση των ε, προτεραιοτήτων της Ευρω... Ρουμανικής Προεδρίας. Ήταν εκτενέστατη η ομιλία σας. Έχουμε 30 ομιλητές που ζήτησαν το λόγο. Γι' αυτό παρακαλώ δύο λεπτά στους συντονιστές και ένα λεπτό στους λοιπούς ευρωβουλευτές. Πρώτος έχει το λόγο ο κύριος ο συντονιστής του ΕΛΚ. Εγώ με διακριτικότητα θα υψώνω το σφυράκι μου όταν πλησιάζεται προς το τέλος του χρόνου. Σας ο κύριος Δέσ. Σε ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε και τον κύριο Υπουργό που ήρθε να μας επισκεφθεί στο Κοινοβούλιο στην Επιτροπή Γεωργίας για να παρουσιάσει το πρόγραμμα της Ρουμανικής Προεδρίας. Αναφέρατε ότι η ΚΑΠ θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην Προεδρία σας. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει πολύ χρόνο στη διάθεσή σας, θεωρείτε ότι θα καταφέρετε να κλείσετε οτιδήποτε. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι εφικτό. Μαζί με τον Παύλο Ντεκάστρο προετοιμάσαμε την διαδικασία που ονομάζεται Omnibus και μας πήρε 14 μήνες. Και ήταν απλούστερη από ότι η ΚΑΠ ως εγχείρημα. Δεν νομίζω λοιπόν ότι η Ρουμανική Προεδρία θα καταφέρει να κλείσει όλα τα θέματα. Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ποιότητα και όχι στην ταχύτητα. Στο τέλος της ομιλίας σας αναφερθήκατε στα δάση. Από την ευρωπαϊκή άποψη τα δάση είναι εθνικός πλούτος, είναι εθνική αρμοδιότητα. Έχουμε 100 εκατομμύρια εκτάρια περισσότερα δάση από ό,τι είχαμε πριν από 30-40 χρόνια. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στα δάση λόγω της ε, αποθήκης αυτά του διοξιδίου του άνθρακα και για διάφορους άλλους λόγους. Αναφέρατε την ανταγωνιστικότητα στο ε, Γεωργία. Ε, σύμφωνα με την πρόταση του Επιτρόπου Χόγκαν, δεν έχουμε ιδιαίτερο περιεχόμενο εκεί. Η ανταγωνιστικότητα προτάθηκαν από τον Επιτροπό Χόγκαν αναφέρατε καλέ ε, τιμέ για τα τρόφιμα. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλέ διαφορε στι τιμέ ε, σε ολόκληρη την Ευρώπη, οπότε θα χρειαστεί να ασχοληθούμε και να συζητήσουμε τα πράγματα κατά χώρα. Δεν πιστεύω ότι οι Βρυξέλλε ε, μπορούν να, να θεσπίσουν όλου του νόμου έγκαιρα. Σα εύχομαι ότι καλύτερο εκ μέρου τους ΕΠΠ. Ο κύριο Καπούτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Πρόεδρο για την έκθεση, για την παρουσίαση, για το περιεχόμενο για τις προτεραιότητε που μας ε, απαρίθμησε ελάχιστα βλέπουμε μια τόσο ολοκληρωμένη παρουσίαση. Πράγματι, όπως λέτε και εσείς, ε, πρέπει να επιταχύνουμε. Έχουμε μπροστά μας ε, στο προσεχές διάστημα φακέλους σημαντικού. Συμφωνώ με τα όσα είπε ο κύριος Ντες όσον αφορά την ΚΑΠ. Οι ενώσεις διαφόρων κλάδων μας ζητούν μια νομική βάση για την επόμενη θητεία. Και εμείς ε, συζητάμε προσπαθώντας να κλείσουμε τις εργασίες στην Κομισιόν ή ε, προσπαθώντας ε, να τις φέρουμε στην Ολομέλεια. Ήθελα να μου πείτε ποια είναι η δική σας άποψη όσον αφορά αυτό. Εσείς αναφερθήκατε σε σχεδόν όλα τα σημεία από τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, αναφέρατε πολλές προτεραιότητες και χαίρομαι που συμφωνώ μαζί σας ε, που αναφέρατε την προτεραιότητα για τους νέους στη Γεωργία. Είναι το θεμελιώδες ε, στοιχείο πιστεύω για τη νέα ΚΑΠ. Θα πρέπει να οικοδομήσουμε μια διαφορετική νέα Γεωργία βάσει της νέας ΚΑΠ. Μια Γεωργία που να μπορεί να καινοτομεί και γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε οπωσδήποτε τους νέους. Η ερώτηση όμως που θέλω να σας απευθύνω είναι διαφορετική. οι γεωργοί θέλουν οι δαπάνε για την ΚΑΠ να βασίζονται, να βασίζονται στου στόχου τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να δείξουμε αυστηρότητα όσον αφορά και τα προϊόντα που μπαίνουν, που εισέρχονται στην Ευρώπη μέσω τη εισαγωγή της υποχρέωσης ε, δήλωση τη καταγωγής ε, στην επισήμανση των τροφίμων. Δεν είναι προστατευτισμός αυτό, ε, δεν είναι παραδιαφάνεια. Μπορείτε να μου πείτε ποια είναι η άποψη τη Ρουμανικής Προεδρία για αυτό το θέμα. Ο κύριο Κουσμιούκ. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω θερμότατα και για την παρουσία σας και για την ε, εκτενή παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Ρουμανικής Προεδρίας. Ε, και όπως και οι προλαλήσαντες, θα ήθελα και εγώ να πω ότι ένα εξάμεινο είναι ελάχιστος ε, καιρός, ελάχιστος χρόνος και σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα έχουμε καν εξάμεινο, θα έχουμε μόνο ένα τρίμηνο, γιατί τέλη Απριλίου θα έχουμε τις τελευταίες μας συνεδριάσεις. Και από αυτήν την άποψη ο χρόνος είναι πραγματικά ελάχιστος. Είπατε ότι μία από τις τέσσερις βασικές σας προτεραιότητες θα είναι η Ευρώπη της σύγκλησης και της συνοχής. Και άρα η μείωση των ανισοτήτων, ο περιορισμός των ανισοτήτων μεταξύ των διαφορών χωρών. Και Ξέρετε, είστε περίπου 12 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς από το 15, ε, εμείς 15 χρόνια και παρόλα αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν τεράστιες διαφορές ε, στις άμεσες ενισχύσεις για τις δικές μας γεωργούς. Και Σίγουρα στο νέο πολιτή δημοσιονομικό πλαίσιο προτείνεται ένα μηχανισμό ε, εξίσωσης των άμεσων ενισχύσεων. Δεν πιστεύετε όμως ότι σε επόμενε δημοσιονομικές προοπτικέ θα πρέπει να έχουμε απόλυτη ευθυγράμμιση, απόλυτη εξίσωση των άμεσων ενισχύσεων. Γιατί ε, αν συνεχιστούν οι ισχύουσες ανισότητες, ε, θα υφίστανται πολύ δυσμενείς διακρίσεις η γεωργοί των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Ερωτώ λοιπόν, η Ρουμανία στη διάρκεια της, της Προεδρίας της θα κάνει κάποια βήματα για μεγαλύτερη εξίσωση, πιο εκτεταμένη εξίσωση των άμεσων ενισχύσεων για όλους τους γεωργούς Ευρωπαϊκής Ένωσης. κυρία Σένερα. Ευχαριστώ πολύ. Στα πλαίσια των προτεραιοτήτων που σχολιάσατε κι εσείς, πιστεύω πως η ΚΑΠ είναι κάτι που μας ανησυχεί ιδιαίτερα όλους. Και θα ήθελα να σας κάνω την εξής ερώτηση. Έχετε σκεφτεί να προωθήσετε κάποια δράση για να υπερασπιστούμε και να δώσουμε προτεραιότητα στις μικρές εκμεταλλεύσεις, στις οικογενειακές, στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ γιατί το συζητάμε συνέχεια, αλλά τελικά ποτέ δεν φτάνουν μπροστά μας προτάσεις για να διατηρηθούν αυτές οι εκμεταλλεύσεις εν ζωή, γιατί αυτές πραγματικά δημιουργούν θέσεις απασχόλησης και επιτρέπουν η γεωργική δραστηριότητα να κρατάει εν ζωή την ύπεθρο. Δεύτερον, γυναίκες. Ρωτώ, νομίζω από τις νέες προτάσεις ΚΑΠ είναι εξαφανισμένες. Θα ήθελα να μου πείτε αν θα προτείνετε εκ μέρους της Προεδρίας κάποιο συγκεκριμένο μέτρο έτσι ώστε να εξαλείψετε τις ανισότητες που επηρεάζουν τις γυναίκες ε, και κυρίως στα πλαίσια των γεωργικών οικογενειακών εκμεταλλεύσεων. Τέλος. Yes. Εμείς έχουμε συζητήσει εδώ στο Κοινοβούλιο, στη δική μας Επιτροπή και έχουμε εγκρίνει και ένα ψήφισμα για την συγκέντρωση γεών στην ε, Ευρώπη. Και σε κάποιες περιοχές, όπως για παράδειγμα η Γαλλικία στην Ισπανία, από την οποία προέρχομαι, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε τεράστιες επιέσεις, αγοράζουν γη μεγάλες επιχειρήσεις και σε πάρα πολλές περιπτώσεις μέσω αυτών των επιχειρήσεων οι οποίες είναι ε, βιομηχανία της γεωργίας, ε, ε, χρησιμοποιούν αυτή τη γη μόνο και μόνο για να θάβουν εκεί τα απόβλητα των χείρων. Έχετε υπόψη να λάβετε κάποια μέτρα έτσι ώστε αυτή η γη να δοθεί σε μικρές επιχειρήσεις. Ευχαριστώ κύριος Χόισλινγκ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε για την παρουσίαση χθες. Ακούσαμε ε, για το ίδιο θέμα στην ε, Επιτροπή ΕΜΒΗ. και θέλω να αναφερθώ στα πράγματα που αναφέρατε και για τα οποία δεν λάβαμε απάντηση χθε στην ΕΜΒΗ για τι μικρέ εκμεταλλεύσει. Αναφερθήκατε εν συντομία. Η Ιρλανδία ε, ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τα συμφέροντα των μικρότερων ε, αγροτών ε, που ασκούν δραστηριότητε διαβίωση. Ε, δεν λάβαμε κάποια απόφαση γι' αυτό. Τι γίνεται με την αρπαγή γεών και αυτό παίζει ρόλο στη χώρα μα. Πρέπει να δούμε πώ θα αντιμετωπιστεί. Πώς θα αντιμετωπίσουμε επίσης την μείωση του πληθυσμού στις γεωργικές περιοχές. Κρίμα που στο δεύτερο πυλώνα ε, υπάρχουν περικοπές για το ζήτημα αυτό. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Επίσης, ε, μου κάνει εντύπωση αυτό που είπατε χθε. Δεν αναφέρατε ε, το κλίμα χθε. Τι σκοπεύετε να κάνετε εσεί και οι υπόλοιποι ώστε να διασφαλίσουμε ότι η Γεωργία θα συμμορφώνεται με τους στόχους καταπολέμησης τη κλιματικής αλλαγής. Θα θέλαμε μια δήλωσή σα και για αυτό το θέμα. Επιπροσθέτω, ήθελα να αναφέρω το εξή Σε ορισμένε, χώρε, όπω και στη δική σα υπάρχουν προβλήματα διαφθοράς. Πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Λείπουν χρήματα τα οποία τα υπεξερούνται διάφοροι. Πρέπει να υιοθετήσουμε τα μέτρα που θα χρειαστούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη διαφθορά. Η χώρα σας ε, δεν κάνει και πολλά για τη μείωση των λιπασμάτων. Δεν είστε και πρωτοπόροι στον τομέα. Εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε ε, αμφίβολα ε, ε, ε, ποιότητα χημικά. Τι να, τι να κάνουμε με μια κάπα αν δεν αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, τα νοικοτινοειδή είναι τα λοιπάσματα στα οποία αναφέρομαι. Υπάρχουν διάφορες οδηγίες ευρωπαϊκές ε, για τα θέματα αυτά και τι γίνεται με την παράνομη υλοτομία. Είναι κάτι που ε, είναι πιο διαδεδομένο στη δική σας χώρα από ότι η, μόνιμη, η νόμιμη υλοτομία. Υπάρχουν προστατευμένες περιοχές τις οποίες ε, είναι αδύνατο να κάνει κανείς υλοτομία χωρίς να ε, παρέμβει η κυβέρνηση. Κάτι πρέπει να γίνει για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Κύριε Σλουαζό, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, η προεδρείς διαδέχονται μία την άλλη και μοιάζουν και πολύ χωρίς να έχουμε θετικές εξελίξεις για τους γεωργούς δυστυχώς. Και αυτό όχι επειδή δεν έχετε αρμοδιότητες ή βούληση, αλλά γιατί όλοι οι προκάτοχοί σας ε, είστε ανίκανοι να εμποδίσετε την επέλαση του ε, βρυξελιώτικου ε, οδοστρωτήρα που ε, καταδυναστεύει τους γεωργούς. Και αυτό είναι το πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ουσιαστικά στηρίζεται στην υποταγή του γεωργικού κλάδου στις ανελαίτες ε, διατάξεις και στους ανελαίτους κανόνες της ε, αγοράς. Και μάλιστα η ΚΑΠ είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αγνοείται τα οικονομικά προβλήματα των γεωργών χωρίς να ξεχνούμε επίσης το γεγονός ότι Δυστυχώ η νέα ΚΑΠ δεν πρόκειται να δώσει ενάψματα για την ανάληψη δραστηριότητα από του νέου γεωργού. Τώρα, ως προς την μεταρρύθμιση. Θα πρέπει να βρούμε λύση πριν το τέλη Φεβρουαρίου για τα τρία σκέλη της ΚΑΠ. δεν θεωρείτε ότι ένα τόσο σημαντικό κείμενο ε, νομοθετικό για τη ζωή των γεωργών θα συζητηθεί σε τόσο λίγο χρόνο. Επίσης, πώς έχει πορεία το συζητήσεων στο Συμβούλιο, ιδιαίτερα για τα θέματα που αφορούν ε, το πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο. Και τέλος, ε, ποιες είναι οι κατευθυντήριες γραμμές για το γεωρικό προϋπολογισμό, ε, είναι, ποιος είναι ο προσανατολισμός της Ρουμανικής Προεδρίας για τις διαπραγματεύσεις του γεωρικού προϋπολογισμού. Ευχαριστώ. Ακούσαμε τους συντονιστές, περνάμε τώρα στις μονόλεπτες παρεμβάσεις. Η κυρία Ζωανάη, αντιπρόεδρος μας. Κύριε Υπουργέ, ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην Επιτροπή μας. Σας γνωρίζω πολύ καλά. Ξέρω πως είστε πάρα πολύ πεπειραμένος και ξέρω πόσο προσπαθείτε έτσι ώστε η γεωργία να είναι στη θέση που πρέπει με πολύ υψηλούς κανόνες και πρότυπα. Και για το λόγο αυτού σας ψήφισαν οι Γεωργοί. Κύριε Υπουργέ, χρειαζόμαστε επικουρικότητα. Αλλά στην Ευρώπη έχουμε ένα πρόβλημα. Φεύγει ο κόσμος από την Ήπεθρο. Θα πρέπει να προσελκύσουμε την νεολαία. Να εμψυχώσουμε τις γυναίκες. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε συγκεκριμένα προγράμματα. Η ψηφιοποίηση εδώ είναι ουσιαστικό. Διαφορετικά η ευρωπαϊκή γεωργία δεν θα σεβαστεί τα πιο απαιτητικά πρότυπα. Εμείς μιλάμε πολύ συχνά εδώ για θέματα όπως ο ενδράση ε, ο ενεργός γεωργός για παράδειγμα, ε, ο νέος γεωργός, ε, Ξέρω πως για το δεύτερο πυλόν εσείς ενδιαφέρεστε πολύ για τις επενδύσεις στα πλαίσια αυτού και τα επενδυτικά σχέδια και αυτό είναι σημαντικό. Τώρα, πιστεύουμε πως χρειάζεται να έχουμε το ίδιο επίπεδο ενισχύσεων για όλα τα κράτη-μέλη και για όλους τους ε, ε, Ευρωπαίους γεωργούς. Τώρα, για το θέμα της ε, ευζοίας των ζώων, να σας πω πως υπάρχουν προβλήματα με το περιβάλλον, αλλά ξέρω παρόλη την παρατήρηση που έκανε ο συνάδελφος πως εσείς το περιβάλλον το σέβεστε ιδιαίτερα. Οπότε το χρόνο που έχω τον ε, διαθέτω ε, στο να σε ευχηθώ καλή επιτυχία και είμαι σίγουρος πως εσείς όταν έχετε με, με εσάς το τιμόνι της, ε, της Ευρωπαϊκής Γεωργίας το θέμα της ΚΑΠ θα τρέξει με θετικά αποτελέσματα για όλους. Η κυρία Ράς Γκαρσία, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ και ευχαριστούμε που ήρθατε. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Είμαι η συγγήτρια της έκθεσης για τα στρατηγικά σχέδια. Ερωτώ λοιπόν, πώς βλέπει το Συμβούλιο την πρόοδο, υπάρχει καταρχήν πρόοδο, σε τι φάση των διαπραγματεύσεων βρίσκεστε, τι πορεία ακολουθεί το Συμβούλιο για το θέμα των στρατηγικών σχεδίων. Επίσης, ε, για το Μερκοσούρ, προβληματίζομαι πολύ με την πρόοδο που μπορούμε να πραγματοποιήσουμε για το Mercosur κυρίω για τι γεωγραφικέ ενδείξει και τι ονομασίε προέλευση. Γιατί κάποιε ονομασίε προέλευση και γεωγραφικέ ενδείξει ευρωπαϊκέ δεν αναγνωρίζεται όπω θα έπρεπε από τι χώρε του Μερκοσούρ. Ποια είναι η γνώμη σα γι' αυτό και ποια είναι τα σχέδια τη Ρουμανική Προεδρία. Και τέλο, για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, θα ήθελα να μου πείτε είναι γεγονό ότι έχουμε και άλλες αναγκαίε ευρωπαϊκές πολιτικές. Για πολλού όμω η μόνη λύση είναι να περικοπούν τα γεωργικά κονδύλια. Για πολλού στο Συμβούλιο εννοώ. Η μόνη λύση είναι να συρρυκνωθεί ο γεωργικός προϋπολογισμός, η ΚΑΠ. Γιατί αντί να συρρυκνώσουμε την ΚΑΠ δεν προτείνεται η ενίσχυση των εθνικών συνεισφορών για το γεωργικό προπολογισμό, κύριε Στουρκάλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσεις για σας. Σας καλωσορίζω φυσικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να σας ε, ρωτήσω όσον αφορά το ανώτατα όρια των επιχορηγήσεων, διότι αυτό παρουσιάζει, η επιβολή τέτοιων ανώτατων ορίων παρουσιάζει και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ποια είναι η δική σας άποψη. όσον αφορά τους ε, κτηνοτρόφους χείρων που αυτή τη στιγμή ε, αντιμετωπίζουν ε, δυσκολίες και όσον αφορά και τους μεγάλους γεωργούς, τα μεγάλα αγροκτήματα. Τι, πώς βλέπετε τις περιοχές, τα αγροκτήματα, τα χειροστάσια. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, συναντηθήκαμε σε μια εκδήλωση της Βουλγαρικής Προεδρίας. Αφορούσε τα διπλά πρότυπα για τα τρόφιμα και ερώτησή μου είναι κατά την Προεδρία σας. Θα ολοκληρωθεί ο τριμερής διάλογος. Όλο συζητάμε για επιφυλάξεις, ε, για αντιευρωπαϊκές δυνάμεις. Αν καταφέρουμε να αποδείξουμε ότι έχουμε ε, χώρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα γλιτώσουμε πολλές ε, ε, συζητήσεις για τα υπέρ και τα κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης ε, για το περίπτωμα των χείρων αφαιρθήκατε ε, και η Τζοάννα μίλησε με τον Περιφερειακό Διευθυντή της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας στη Ρουμανία. Ο Περιφερειακός Διευθυντής εστάλει στο Ρούσιο όπου την περασμένη εβδομάδα εγώ οργάνωσα μια διάσκεψη και η ερώτηση μου είναι η εξής. Θα ήσασταν υπέρ της χρηματοδότησης. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου, ε, δώστε μου λίγο χρόνο. Ε, μου κάνει έκπληξη ότι με τη νέα Προεδρία αυτή, ξέρω ότι είμαστε πολλοί, μας δίνετε μόλις ένα λεπτό για προβλήματα ύψης της σημασίας. Είτε μιλάμε για τη μελλοντική ΚΑΠ, είτε για τα προβλήματα που ανέφερε ο κύριος ε, Πρόεδρος. Δεν θα σας θέσω πολλές ερωτήσεις όπως συνάδελφοι, πολλές τις έχουν κάνει ήδη. Αλλά θέλω να σας πω κάποιες σκέψεις. Ως βουλευτής ε, ε, είμαι εξωφρενών με τις απειλές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απειλούν μετά την Ουγγαρία και την Πολωνία και εσάς τώρα απειλούν για αποτρεπτικά περικόπτοντας κομμάτων ε, ενισχύσεων που θα δοθούν σε εσά. Σε μια χώρα που η δική σας, ε, άκουσα και τους μικρούς γεωργούς ε, απελπισμένους λόγω της πίεση των πολυεθνικών που έχουν καταλάβει τις καλύτερες γεές σε φθηνέ τιμές και έτσι λαμβάνουν τις περισσότερες επιχορηγήσεις. Στη Βουλγαρία οι άμεσες ευρωπαϊκές ενισχύσεις στους μικρούς γεωργούς αφορούν λιγότερο από το 10% αυτών. Όσον αφορά τη δική σας χώρα, εμείς υποστηρίζουμε τις πολιτικές ε, που επιτρέπουν στους Ρουμάνους ε, εργαζομένους να επανέρχονται στη χώρα τους αντί να αποτελούν το αντικείμενο εκμετάλλευση από πολυεθνικές ε, στο πλαίσιο της απόσπασης εργαζομένων σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, σε τέτοιες εποχές αγροτικής κρίσης και διεθνών εντάσεων, συμφωνώ και μαζί σας και θέλω να σας επιστήσω την προσοχή όσον αφορά την προσέγγισή σας με τους ε, ανατολικούς σας ε, γείτονες. Η Μολδαβία ε, τότε που επιβλήθηκε το ρωσικό εμπάργο είχαν την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δυνατότητα εξαγωγής των ε, δικών των γεωργικών παραγωγών χωρίς δασμούς. Αυτό επηρέασε τους δικούς μας παραγωγούς και επηρέασε και τις εμπορικές συνθήκες. Ε, εξαγωγής προϊόντων από την Ουκρανία στην Ευρώπη. Μετά η χρήση της γεωργίας ε, ως ε, διπλωματικού εργαλείου δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα πολλών πολιτών των κρατών μας με δραματικές συνέπειες. Έχει έρθει η ώρα να φτάσουμε σε μια πιο λογική προσέγγιση που θα ευνοεί περισσότερο του γεωργού των χωρών μα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα κι εγώ να επαναλάβω όσα είπαν οι συνάδελφοι, κυρίως για το χρονοδιάγραμμα. Είναι ρεαλιστικό. Δεν νομίζω. Πολλοί από τους ευρωβουλευτές δεν το πιστεύουν και αυτό ανεξάρτητα της πολιτικής ομάδας. Μία ακόμα ερώτηση. Τι νομίζετε και πώς, απο... και πώς αντιμετωπίζετε την ε, απόφαση της Κομισιόν για τις οροφές, γιατί πάρα πολλοί είπαν πως είναι παράλογο και αρκετοί προσπαθούν η ΚΑΠ να γίνει πιο αξιόπιστη. Εγώ είμαι και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμών και πρέπει να σας πω πως από τότε που είμαι εκεί πάρα πολλοί φωνάζουν πως κάτι χρειάζεται να αλλάξει. Φαίνεται όμως πως όταν φώναζαν δεν τους άκουγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι πιστεύετε, θεωρείτε κι εσείς πως στερείται νοήματος αυτή η προσπάθεια επιβολής οροφών. Κύριε Σαντρία, ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ που ήρθατε και καλώς ήρθατε. Το θέμα της αστάθειας των τιμών και της σταθερότητας των αγορών είναι πολύ σημαντικά για το μέλλον της γεωργίας, γιατί ε, υπονομεύει όλο τον κλάδο. Το συζητήσαμε και στα πλαίσια της ΚΟΑ, της Κοινή Οργάνωσης Αγοράς της Μελλοντικής Μεταρρύθμισης. Και φαίνεται ότι υπάρχει βούληση να γίνει η ΚΟΑ εργαλείο πρόληψη ε, η διαχείριση των κρίσεων, δίνοντα περισσότερε ευθύνε στην Επιτροπή για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των κρίσεων. Αυτό όμω προποθέτει μεγαλύτερη διαφάνεια. Επίσης, ε, ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σα. Ε, πιστεύετε ότι η κοινή οργάνωση αγορά μπορεί να γίνει διαχειριστικό εργαλείο, εργαλείο διαχείριση των αγορών. Και μάλιστα με βάση τι εργασίε για τον κανονισμό Omnibus, φαίνεται η προσπάθεια ενίσχυσης της οργάνωση των γεωργών σε οργανώσεις και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών. Στα πλαίσια της ε, δικής σας προεδρίας και παρά το ελάχιστο χρονικό διάστημα που θα έχετε, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε πολλές διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική μεταρρύθμιση της ΚΑΠ δεδομένου του χρονοδιαγράμματος. Πώς θα προωθήσετε αυτές τις ιδέες για την καλύτερη οργάνωση των παραγωγών και επίσης για τη διαφάνεια των αγορών. Τι θα προτείνετε στο Συμβούλιο. Ε, είναι περίπλοκη η κατάσταση και ελάχιστος ο χρόνος. Ποιες βλέπετε να είναι οι συνέπειες του Brexit στη Γεωργία, κυρίως στο εγγύς μέλλον. Ευχαριστώ. Ε, κυρία Κλονέκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Έλειψα λίγο όταν πήρατε το λόγο, αλλά μιλήσατε για τα πρωτεϊνούχα φυτά και ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας καλωσορίσω και εγώ στην Προεδρία. Ξέρετε και εσύ πως 22 Νοεμβρίου πέρυσι η Κομισιόν παρουσίασε μία ε, ε μελέτη, μία έκθεση ε, για τα πρωτεϊνούχα φυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την καλλιέργεια αυτών που είναι απογοητευτική γιατί δεν προσφέρει ένα όραμα για το συγκεκριμένο θόμα τουλάχιστον στα πλαίσια της μελλοντική μεταρρύθμισης της ΚΑΠ. Στην έκθεση αυτή λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει πως η κατάσταση είναι ανησυχητική. Γιατί? Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει ακατέργαση 17 εκατομμύρια τόνους ε, πρωτεϊνούχων φυτών, ε, εκ των οποίων οι 13 είναι υποπροϊόν σόγιας. Και παράλληλα αυτή τη στιγμή διαπραγματευόμαστε με τις ίπα έτσι ώστε να κάνουμε εισαγωγές ακόμα μεγαλύτερες από σόγια στα πλαίσια ε, μιας βιωσιμότητας η οποία αυτή τη στιγμή δεν περιγράφεται. Πείτε μου λοιπόν στα σχέδιά σας τι θα κάνετε, θα αναλάβετε δράση έτσι ώστε ε, να αντιμετωπίσετε αυτή την ε, ε, αντιφατική στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Ερντός. Σύμφωνα με τις πρόσφατες ειδήσεις που διαβάζουμε στον τύπο, Πρόσφατα βρέθηκαν ε, τρόφιμα χειρότερη ποιότητα στι χώρε τη Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Ελέγχεται λοιπόν αποτελέσματα όσον αφορά τη διαφορά ποιότητα μεταξύ Ανατολική και Δυτικής Ευρώπη και την καταπολέμηση αυτού του προβλήματο. Σε ένα ψήφισμα το Κοινοβούλιο πέρυσι ζήτησε να, να απαγορευτούν τέτοιε πρακτικέ. Εσεί ε, συμφωνείτε. Το θέμα αυτό συζητήθηκε ε, σκοπεύετε να το συζητήσετε και εσείς ε, στην Προεδρία σας. Μετά και το θέμα της ε, Αφρικανικής Πανόλης των Χείρων που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ίσως θα πρέπει να αυξηθούν οι πόροι που θα βοηθήσουν ε, τους κτηνοτρόφους ή θα τους αποζημιώνουν. Συμφωνείτε εσείς με αυτό. Ευχαριστώ. Καλημέρα, Πρόεδρε. Ευχαριστώ ε, συναντηθήκαμε χθε στην Επιτροπή Περιβάλλοντο. Δεν θα επαναλάβω τα όσα είπε ο συνάδελφο Ανδρέα για τι ασταθεί τιμέ και την ανάγκη υλοποίηση των εργαλείων διαχείριση κρίσεων. Πρέπει να υλοποιήσουμε και εργαλεία διαχείριση ε, κινδύνου. Διότι περί αυτού πρόκειται σήμερα. Αυτή η ΚΑΠ, η κοινή αγροτική πολιτική, πρέπει να παραμείνει κοινή. Η πρόταση της Κομισιόν δείχνει διάφορες άλλες οδούς ε, επανεθνικοποίησης, ε, επανακρατικοποίησης. Θέλω να αναφερθώ σε ένα ζήτημα. Αναφερθήκατε στη βιοοικονομία. Ε, αυτή τη στιγμή αναθεωρείται ένα κανονισμό. Αναμένουμε τι κατεξοδότηση πράξη, στον οποίο θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σα, διότι είναι σημαντικό για του παραγωγού βιοκαυσίμων που παράγουν και ζωοτροφές όπως ανέφερε ο συνάδελφος μόλις τώρα ε, πρωτεϊνούχες ζωοτροφέ, μιλάμε για την ε, πρόκειται για την αναθεώρηση 2 η ΡΕΒ 2 προσέξτε να μην στραφεί αυτή η οδηγία κατά των Ευρωπαίων γεωργών μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα αλλά θα πρέπει να συνεχίσει να του προστατεύει, να του προστατεύει από τι εισαγωγέ και κυρίω αυτέ του grazie. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Υπουργό και να ευχαριστήσω και την ομάδα της Ρουμανικής Προεδρίας για την υποστήριξη που προσέφεραν μαζί με την Αυστριακή Προεδρία για να ολοκληρωθεί η πολιτική συμφωνία της 19ης Δεκεμβρίου για τις ε, αθέμητες πρακτικές. Εμείς καλούμαστε σήμερα μετά από αυτή την ε, συζήτηση και την ψηφοφορία, οπότε πιστεύω θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε γρήγορα ε, προγραμματίζοντας την ψηφοφορία στην Ολομέλεια στην επόμενη, ε, στην πρώτη του Μαρτίου. Δεδομένων αυτών για την ΚΑΠ, ήθελα να κάνω μια ερώτηση, κύριε Υπουργέ. Δεδομένων των ανησυχιών που ακούμε συχνά στην Επιτροπή μας και δεδομένης και της έκθεσης που ψηφίσαμε του συναδέλφου Ντόρφμαν με μεγάλη συντριπτική πλειοψηφία, μας ανησυχεί που αυτή η πρόταση μεταρρύθμισης θα μπορούσε να οδηγήσει σε κίνδυνο επανακρατικοποίηση. Εσείς ως Ρωμανική Προεδρία τι άποψη έχετε για αυτό το σημείο όσον αφορά τη γεωργική πολιτική. Κύριε Ροπέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ. Άκουσα με μεγάλη προσοχή την ομιλία σας και διαπίστωσα ότι είστε εξοικειωμένο ε, με την κατάσταση τη Γεωργία και στη Ρουμανία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα εύχομαι καλή επιτυχία. Χαίρομαι που προτεραιότητά σα είναι και η σύγκληση. Και κάτι που ρώτησαν και οι συνάδελφοι, με προβληματίζει και εμένα. Τι επίπεδο σύγκληση θα επιδιώξετε, Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μίλησε για μείωση κατά 50% των ανισοτήτων. Αλλά οι χώρες της Βαλτικής και η γεωργοί της Λιθουανίας έχουν μεγαλύτερες φιλοδοξίες και προσδοκίες από εσά. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ένα αξιοπρεπές γεωργικό εισόδημα και η άμεση ενισχύση είναι μόνο το 25% του συνολικού του εισοδήματος. Το υπόλοιπο προέρχεται από τις τιμές των γεωργικών προϊόντων. Πώς λοιπόν σκοπεύετε να προτείνετε σε ένα, ένα μηχανισμό που θα εξασφαλίσει αξιοπρεπείς αμοιβέ για τους γεωργούς ο κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που ήρθατε. Σας εύχομαι καλή τύχη και καλή επιτυχία στην Προεδρία σας. Θα ήθελα να μιλήσω για την αρπαγή των γεών, ιδιαίτερα στην Ανατολική Ευρώπη. Δεν ξέρω αν με ακούτε κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση η, η αρπαγή των γεών στην Ανατολική Ευρώπη είναι ένα εκτεταμένο φαινόμενο, ένα πολύ ε, γενικό φαινόμενο στην Γερμανία, στην Ανατολική, στην Ανατολική Γερμανία, στη Ρουμανία και σε άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Ποια είναι η γνώμη σας για το φαινόμενο αυτό, δεδομένου ότι οι ευρωπαϊκές γεωργικές επιδοτήσεις πολύ συχνά καταλήγουν στα χέρια κερδοσκόπων που μερικές φορές δεν είναι καν ε, ε κοινοτική, είναι ε, εξοκοινοτική. Σε ό,τι αφορά την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων, ε, μπορείτε να μας ενημερώσετε για το βαθμό μετάδοσης της επιζωτίας αυτής στη Ρουμανία, σε ό,τι αφορά τη μικροβιακή αντοχή. Πώς βλέπετε την πιθανότητα μόλυνσης από τα κτηνιατρικά φάρμακα γιατί δεν ξέρουμε ποιος είναι ο φορέας αυτής της έκτασης, εξάπτωσης. Όταν, πήγε, η, όταν μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ρουμανία είχαν μια πολύ στεναρή βιομηχανία ε, παραγωγής ε, γενετικά τροποποιημένης σόγιας και ερχόντουσαν Γεωργοί ε, σε μένα με φωτογραφίες και μου λέγαν κοιτάξτε τις καλλιέργειες μου ε, όταν είναι γενετικά τροποποιημένη η σόγια είναι ε, τα βλαστάρια τρυφερά και τα υπόλοιπα κοιτάξτε τις φωτογραφίες είναι χάλια και παρόλα αυτά τους είπα σταματήστε. Σταματήστε δεν χρειάζεται πια γιατί δεν επιτρέπεται. Οπότε αφήστε στην άκρη τα δάση δεν είναι ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Αφήστε ε, το κλίμα στην άκρη, δεν φταίνει η γεωργία για το κλίμα στον κόσμο και κάντε αυτό που είπατε, ε, αντιμικροβιακή ανθεκτικότητα. Αυτό πρέπει να το επιδιώξουμε και εκεί οι γεωργοί μπορούν να δώσουν πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω κύριε Υπουργέ, γιατί είχαμε τη δυνατότητα και στην Αλία να σας ακούσουμε, τώρα και στη Γεωργία, να σα πω πως χρόνος υπάρχει λίγος. Και ήθελα και εγώ να συνταχθώ με του συναδέλφους. Δεν έχουμε χρόνο για να κάνουμε μια μεταρρύθμιση τη κάψαν αυτή που περιγράφουμε. Και επίση θα ήθελα, και το είπε ήδη ο Παόλο Ντεκάστρο, να μου πείτε τι θέλει η κυβέρνησή σας και πώς αντιμετωπίζει την ε, πρόταση με τα εθνικά στρατηγικά σχέδια ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που για μας είναι ε, επεθνικοποίηση της ΚΑΠ και τι θα κάνουν, θα αναλάβουν τα ενία της Γεωργίας πια τα κράτη-μέλη και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχούμε, δεν υπάρχει χρόνος και νομίζω πω πως αυτή τη θητεία δεν θα προλάβουμε. Επίσης, να σας πω πως είναι σημαντικό να δώσετε τη μάχη για καλό προϋπολογισμό, να έχουμε τον προϋπολογισμό στα ύψη που ήταν στο παρελθόν και όταν έρθει η συζήτηση ε, για, τις για, τα... για το πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο, να καταλάβετε πως τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά κάπου χρειάζεται χρήματα. Και τουλάχιστον να μείνουμε στα σημερινά επίπεδα. Κύριε Σβάιτς. Äh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αναφερθήκατε σε ειδικέ διατάξεις για τα νεονικοτινοειδή. Τι θα γίνει με αυτό το μέτρο έκτακτη ανάγκη, ποια είναι η στρατηγική σας εδώ. Αξιολογήθηκε ε, στο πλαίσιο της ελαιοκράμβης Γιατί τι βλέπετε με το καλαμπόκι και το... Τι θα γίνει με το μείωση του γεωργικού προπολογισμού στο σύνολό του, ειδικότερα στο πλαίσιο του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου που ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, θεωρείτε ότι ο προπολογισμό για τη γεωργία θα πρέπει να μειωθεί ή ότι όχι, ή συμφωνείτε με το πρόγραμμα εξοικονόμηση τη Κομισιόν. Κύριε Χόιμπουχ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, είπατε ότι η κοινή γεωρική πολιτική θα πρέπει να προσαρμόζεται και στις μελλοντικές προκλήσεις, ε, τις κλιματικές, τις περιβαλλοντικές. Εγώ διαφωνώ με τον κύριο Άγνιο ότι θα πρέπει να αφαιρέσουμε τους κλιματικούς μας στόχους από τη γεωργία. Γιατί αλλιώς ε, τις αρνητικές συνέπειες των κλιματικών αλλαγών θα τις υποστούν κυρίως η Γεωργία. Επίσης, ε, τι πολιτική θα προτείνετε στο Συμβούλιο για τις αγορές. Υπάρχει τεράστια αστάθεια στις τιμές και είναι με την πλάτη στον τοίχο η Γεωργή. Επίσης, ε, είπαμε ότι θα πρέπει κάπου να στηρίζεται στις ευρωπαϊκές συνθήκες και θα πρέπει οι υπόλοιπε πολιτικές μας να είναι ε, συναφείς ε, με την αναπτυξιακή μας πολιτική. Βέβαια, η γεωρική πολιτική επηρεάζεται και από πολλού εξωτερικού παράγοντε. Γι' αυτό θα ήθελα να σε απευθύνω έκκληση να εξασφαλίσετε μια πολιτική συνοχή και τη κοινή γεωρικής πολιτική και συνοχή και συνάφεια με τι υπόλοιπε μα πολιτικέ για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Και μάλιστα το συζητήσαμε αυτό ιδιαίτερα στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Κύριος Μπόκοβιτς. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ που είστε μαζί μας σήμερα. Σας εύχομαι καλή τύχη για την Προεδρία σας και έχω δύο ερωτήσεις να σας κάνω. Πρώτον, η ε, συνένωση μεγάλων εκμεταλλεύσεων άνω των χιλίων εκταρίων είναι ένα τεράστιο πρόβλημα στην Ευρώπη. Η οικογενειακή γεωργία βρίσκεται υπό απειλή εξαιτία αυτών. Στην πρόταση κανονισμού ε, του στρατηγικού κανονισμού προβλέπεται μείωση των πόρων για το σκοπό αυτό από 60.000 ε, και από τις 100.000 να καταργούνται τελείως. Δεύτερη ερώτηση, η πρωτοβουλία του εφιούς χωριού με σκοπό τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και των δραστηριοτήτων στις γεωργικές περιοχές ε, για, από κοινωνική άποψη τα ε, νηπιαγωγεία, τους παιδικούς σταθμούς, ε, ό,τι χρειάζεται για να μένουν οι νέοι στις γεωργικές περιοχές. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Ποιες είναι οι προθέσεις σας, οι θέσεις σας επί του θέματος και θα λάβετε υπόψη όλα αυτά τα θέματα. Κύριε Πετήρ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τον Προεδρεύοντα για την παρουσία του. Η Γεωργία ε, θα αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα και έχει πολλές προκλήσεις και όσα βήματα προόδου και αν κάνουμε, δύσκολο, δύσκολα θα ανταποκριθούμε άμεσα σε όλες τις ανάγκες των γεωργών. Και θέλουμε μια ηλικιακή ανανέωση, όπως είπατε. Θέλουμε νέους γεωργούς στη γεωργία. θα πρέπει να μας ακούσει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τα 50.000 αν έλθει στα 100.000 ευρώ. Και επίσης ε, ε, αυτό ήταν ε, ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την πρόσληψη νέων. Ελπίζω να μας ακούσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να λάβει υπόψη τις προτάσεις μας για να έχουμε την ηλικία και ανανέωση. Επίσης, να μιλήσω για μια ομάδα που είναι τελείως παραμελημένη όταν μιλούμε για την ανάπτυξη υπαίθρου. Μιλώ για τις αγρότησες, για τις γυναίκες στην υπαίθρο. Και έχουμε μεγάλο ποσοστό οικογενειακών εκμεταλλεύσεων και από το 2014 το 35% του χρόνου τους ε, το αφιέρωσαν στην ε, γεωργική δραστηριότητα και ταυτόχρονα ε, ασχολούνται με την οικογένειά τους, φροντίζουν τα παιδιά τους, ανατρέφουν τα παιδιά τους και παρόλα αυτά η εργασία τους δεν αναγνωρίζεται. Αγνοείται πλήρως. Τι γνώμη έχετε για τις αγρότησες, για τη γυναίκα στην Ήπεθρο, γιατί πραγματικά είναι πολυδιάστατο το έργο του και χάρη σε αυτές σε μεγάλο βαθμό εξασφαλίζεται η επιβίωση στην Ήπεθρο. Κύριε κυρία Μαγκίνες. Ακούστηκαν πάρα πολλέ συζητήσει πρόσφατα για το θέμα της υγείας και της διατροφής και το κλίμα και στην έκθεση αυτή πρέπει να σα πω ότι ε, σχολιάσαμε θέματα, όλα συζητήθηκαν, αλλά μιλήσαμε για την εντικοποίηση της παραγωγής με βιώσιμο τρόπο στην υφιστάμενη γη. Πιστεύετε πως η ΚΑΠ θα βοηθήσει προ αυτή την κατεύθυνση? Και θα ήθελα να μου πείτε με ποιο τρόπο γιατί οι παραγωγοί ανησυχούν ιδιαίτερα για αυτά τα μεικτά μηνύματα τα οποία λαμβάνουν από χαράσουν πολιτική και σε παγκόσμιο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ανησυχούν για το κατά πόσο τα εισοδήματά τους θα είναι βιώσιμα και αν θα είναι και οι εκμεταλλεύσεις τους ε, βιώσιμες. Οπότε ναι, θα γίνει αυτή η νέα γεωργική επανάσταση στην Ευρώπη γιατί αυτή πρότεινε η Επιτροπή, η έκθεση Λάντσφερτ και τελικά ε, περιορίστηκε σε θέματα διατροφής. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Στην Ευρώπη μερικές φορές για εβδομάδες και ολόκληρες μεταφέρονται ζώα και υποφέρουν τρομακτικά. Μ' αρέσει που έχετε βάλει ω προτεραιότητα να αλλάξει αυτή η κατάσταση ω Ρουμανική Προεδρία. Θέλω να αναφερθώ στην έκθεση για την εφαρμογή των νέων κανόνων, όπου ζητείται περιορισμό των μεταφορών αυτών αριθμητικά και απόψη διάρκεια. Συζητείται επίση και μείωση των μεταφορών προ τη Μέση Ανατολή. Αντί όμω να ακούει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ρουμανία κάνει το αντίθετο είναι ο κύριος εξαγωγός ε, ζωντανών ε, προβάτων. Μάλιστα, έχετε συνάψει συμφωνίες ε, με την Αρμαβασή, μια εταιρεία μεταφορική που μεταφέρει για λογαριασμό σας τα ζώα προς άλλες χώρες πάρα πολλά εκατομμύρια ζώα είναι το αντικείμενο αυτών των, αναφορών, των μεταφορών. Για παράδειγμα, η Αυστραλία, ξέρετε, έχει διακόψει κάθε επαφή με αυτή την επιχείρηση. Εσείς όμως Πώς το βλέπετε, τι θα κάνετε, ε, πώς, μπορείτε να συνάπτετε ε, συμβάσεις με μια τόσο αμφίβολη ποιότητα εταιρεία, πώς θα διασφαλίσετε την καλή μεταχείριση των ζώων, κάτι που σας ζητά και σας απαιτεί μεγάλη συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωπαίων. Ευχαριστώ, δεν υπάρχουν άλλοι ε, εγγεγραμμένοι. Έχουμε ολοκληρώσει τις ερωτήσεις πολύ ε, παρενέβησαν ε, πολλές ερωτήσεις. Να ζητήσω από τον Υπουργό τώρα να απαντήσει στις ερωτήσεις. Δεν σας επιβάλλουμε κάποιο χρόνο, αλλά μπορείτε να είστε σύντομος. Ε, παρακαλώ κύριε Υπουργέ. Μα Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος, αν μπορώ. Αλλά τα ζητήματα είναι μεγάλα Χθε βρέθηκα στην Επιτροπή Ένβη. Και εκεί συζητήθηκε η ΚΑΠ. Και εκεί άκουσα πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις. Όπως και σήμερα στην Επιτροπή Αλίας. Όπου άκουσα ερωτήσεις ε, σαν τις δικές σας. Εγώ χαίρομαι που μου κάνουν ερωτήσεις ε, ε, για θέματα τα οποία που μας αφορούν κάτι το οποίο έχουμε ήδη και θέλουμε να βελτιώσουμε βάσει των όσων έχουμε ήδη και βάσει και προτάσεων της Κομισιόν. Κατά τη δική μου άποψη, η κοινή γεωργική πολιτική ως έννοια βασίζεται ε, στο επίκεντρο της ανθρώπινης ε, ε, ζωής. Έτσι πρέπει να τη βλέπουμε και έτσι πρέπει να την υλοποιούμε. Στις ερωτήσεις που τέθηκαν Αντιληφθήκα ότι εκφράζεται πολλοί από εσά ανησυχίε ε, για πολύ περίπλοκους τομεί. Σας είμαι ευγνώμων λοιπόν για όλες αυτές τις ερωτήσεις. Διότι με εμπνέουν να προωθήσω αυτή τη διαδικασία λήψη αποφάσεων προ όφελο των Ευρωπαίων αγροτών και όχι μόνο αυτών. Ε, θα πρέπει όμως να ξεχωρίσουμε κάποια πράγματα να... από κάποια άλλα. Το Νοέμβριο του 2017 η Κομισιόν δημοσίευσε το νέο της ε, μοντέλο για την ΚΑΠ. Και τώρα στις Βρυξέλλες, ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο εμείς ε, σχεδιάζουμε την αρχιτεκτονική μιας πολιτικής που θα φέρει τα όποια αποτελέσματα φέρει το 2021-2027 έως το 2027. Βάσει των όσων θα θεσπίσουμε, εμεί χρειαζόμαστε ένα σαφέ νομικό πλαίσιο ώστε να έχουμε στα χέρια μας τα απαραίτητα εργαλεία για την περίοδο 2021-2027. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε σκεφτεί μεταβολή της ε, όλης έννοιας, αλλαγής της ε, κατά τρόπο ουσιαστικό βάσει μιας επιθυμίας βελτίωσης της κοινή ε, γεωργικής πολιτικής για να καλύπτει τις σημερινές ανάγκες και τις πιθανές μελλοντικές ανάγκες. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ τώρα σε διάφορα από αυτά τα σημεία, ελπίζοντας ότι θα καταφέρω να απαντήσω ικανοποιητικά τι ερωτήσει σα. Ήταν τόσε πολλέ. Ε, και ο χρόνος δεν αρκεί για να μπορέσω να τα πω όλα. Όλοι μας ε, είπαμε ότι θέλουμε απλούστευση της γεωργικής πολιτικής. Από όσο γνωρίζω, από τους γεωργούς της Ρουμανίας και τους γεωργούς άλλων χωρών στο Συμβούλιο με εκφράζεται επιθυμία για μεγαλύτερη επικουρικότητα. Όχι για επανακρατικοποίηση της ΚΑΠ. Διότι Α, απαιτείται να γίνει κάποια αλλαγή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, λάβει τα μέτρα για να γίνουν απαραίτητε αλλαγέ. Και εμείς από τις αντιδράσεις των Υπουργών θα δούμε ποιες είναι οι θέσεις των κρατών. Που ουσιαστικά αποτυπώνουν τα συμφέροντα των αγροτών στα εκάστοτε κράτη-μέλη. Ανέφερα τους πέντε κανονισμούς που χρήζουν τροποποίησης. Έχουμε το στρατηγικό σχέδιο, η χρηματοδότηση, η διαχείριση, εξυγχρονισμός και η κοινή οργάνωση αγορών. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην οργάνωση των εργασιών μας και στη λήψη αποφάσεων και πραγματικά ο χρόνος δεν είναι δεν είναι πολλοί. Το, το έχω πει και εγώ. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο πρέπει να καθίσουμε όλοι μαζί και να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα ώστε τα πράγματα να μπουν σε μια τροχιά. Το είπα καθαρά, έτσι πιστεύω, ότι η ΚΑΠ ε, δεν είναι απλά η ΚΑΠ. Αλλά ε, ε, τι επίπεδο θα έχει η ΚΑΠ στο μέλλον. όπως αποφασίζεται στο Συμβούλιο. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να κάνουμε τις προκαταρκτικές εργασίες καλά, να φτιάξουμε σωστά θεμέλια, σωστές βάσεις. Να καταφέρουμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας, ώστε να βρεθούμε σε μια θέση όπου θα μπορέσουμε να κινήσουμε τα πράγματα κάπως, διότι όλοι είμαστε ε, αλληλένδετοι. Μπορεί να διαφέρουν οι απόψεις μας, μπορεί να διαφέρουν οι ερμηνείες μας, αυτό δεν είναι παράλογο. Γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταφέρει να, επιτύχει μεγαλύτερο βαθμό ελευθερία μέσα των εθνικών στρατηγικών σχεδίων, ούτω ώστε τα επιμέρου κράτη-μέλη να μπορούν να λαμβάνουν ε, υπόψη καλύτερα τα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είτε μιλάμε για το μέγεθος των αγροκτημάτων, είτε μιλάμε για την τοπογραφία ε, της χώρας. Τα κράτη-μέλη είναι εκείνα που φυσιολογικά κάνουν αυτά τα πράγματα που θα μπορέσουν να ε, εκπονήσουν τις απαραίτητες ε, δράσεις και συνέργειες. Διότι αφενός πρέπει να ανήκει κανείς στον δρόμο για τις νέες γενιές Το 34% των γυναικών, για παράδειγμα, που έχουν κάποιο όραμα για αυτό το κλάδο, πρέπει να υποστηριχθούν, να αναφέρονται σαφώς ε, σε ένα νομικό εργαλείο, το οποίο θα χρησιμεύσει όλους μας. Γι' αυτό το λόγο η κλιματική αλλαγή Το είπα και χθε ε, στην ΕΜΒΗ. Και σήμερα στην Αλία μίλησα για τη θάλασσα και τώρα ήρθα εδώ για να μιλήσω για τη γη. Τη γη όπου θέλουμε να καλλιεργούμε αλλά όπου επηρεάζεται σαφώς και το περιβάλλον, οπότε πρέπει οι καλλιέργειες να γίνονται με έναν τρόπο ισόρροπο. Ακούσαμε ερωτήσεις. Έγιναν ερωτήσεις για τη χρήση των λιπασμάτων, των φυτοφαρμάκων. Ε, εντάξει, θεμητό. Αλλά οι γεωργοί χρειάζονται και εναλλακτικέ. εναλλακτικά προϊόντα τα οποία να μπορούν να χρησιμοποιήσουν ώστε να συνεχίσουν να παράγουν, να μπορούν να καλύψουν τις διατροφικές ανάγκες και να μπορέσουν ε, να κερδίζουν και τα προστοζήν. Να μπορούν να επιβιώσουν βάσει των, ε, από τις γεωργικές δραστηριότητε. Να είναι η γεωργία που ασκούν βιώσιμη, να είναι πραγματικοί αγρότες. Που αφενός ε, να μπορούν να παράγουν Αυτό που σχεδιάζει ο ε, γεωπόνος και ε, προγραμματίζει ο οικονομολόγος. Ε, ξέρετε, έχουν υποθεί πολλά για την κλειφωσάτη. Για να τερμινεύσω όλα αυτά βάσει της δικής μου εμπειρίας ε, που είναι μακρόχρονη ως ειδικό σε γεωργικά θέματα. η Η παράταση της χρήσης της γλυφοσάτη για μία ακόμη πενταετία έχει νόημα. Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι τα ζυζάνια αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα από τα υπόλοιπα φυτά. Έχουν ε, άλλη φυσιολογία και είναι δύσκολο να ελέγξουμε αυτά τα ζυζάνια αν δεν έχουμε φυτοφάρμακα που τα χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να εξολοθρεύσουμε τα ζυζάνια. Γι' αυτό λοιπόν είναι απαραίτητο να βρούμε μια ισορροπία. Μια ισορροπία που προσδιορίζεται αφενός από τις δυνατότητες που έχει ο κάθε γεωργός και αφετέρου από το νομοθετικό πλαίσιο που έχουμε δημιουργήσει εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μια παρακολούθηση των καλλιεργειών. Ε, μου θέσετε μια ερώτηση για τα νεονικοτινοειδή. Αυτό όντω είναι πρόβλημα για πολλές χώρες. Η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Φιλανδία, η Εστονία, η Λιθουανία αντιμετωπίζουν τέτοιο πρόβλημα. Και ε, στο χώρο αυτό που έχουμε για το τανιμέκους λατικόρης και για άλλα φυτά ατικόρης ή ποικιλίε ε, φιλοξήρας ή φιλοτέρες για τα ξυλώδη πόδι. Έχουμε πολύ σημαντικές ποικιλίε για το, για το καθημερινό έργο του Γιώργου και ανάλογα με, τη σπορά που, με, τα, με τους σπόρους που έχει χρησιμοποιήσει επιλέγει και το φυτοφάρμακο που θεωρεί κατάλληλο. Ε, και φυσικά προτιμά τα λιγότερο προβληματικά για το περιβάλλον φυτοφάρμακα και τα λιγότερο δαπανηρά. Ο πρόεδρος προσπαθεί να με διακόψει, αλλά θα συνεχίσω για λίγο ακόμη. Μην ξεχνάτε ότι στην αρχή παρακολούθησα και την εσωτερική σας συζήτηση, κάτι που καθυστέρησε τη δική μου ανταλλαγή απόψεων. Και θα ήθελα να σας πω ότι τρέφω ιδιαίτερο σεβασμό προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο και προς τους Ευρωβουλευτές, γι' αυτό και θα βάλω μια τελεία και μια και έχουν μείνει αναπάντητε ερωτήσεις, θα σας στείλω γραπτός απαντήσεις, ώστε να μπορέσετε και εσεί να αξιοποιήσετε το χρόνο σας καλύτερα και να μην σας κουράζω εδώ. Με την ανάγκη μου να μακρηγορήσω. Θα σταματήσω λοιπόν εδώ. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Και Ελπίζω να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα θέματα της συναπόφασης, γιατί μας ενδιαφέρει η νέα κυνηγιορική πολιτική για την περίοδο 2021-2027. Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Υπουργέ, γιατί ήσταν πολύ διεξοδικός και στις απαντήσεις και στην αρχική σας ομιλία και δώσατε πολλές απαντήσεις γιατί όντως το θέμα είναι πολύ πλούσιο και προσφέρεται για εκτενή συζήτηση και εσείς είστε ιδιαίτερα πεπειραμένος στα γεωργικά ζητήματα. Γι' αυτό θα μπορούσαμε να παρατείνουμε πολύ περισσότερο στην την ανταλλαγή απόψεων, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε αρκετό χρόνο. Γι' αυτό πρέπει να ολοκληρώσουμε εδώ αυτό το θέμα και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία σε αυτή τη δύσκολη προεδρία που θα έχετε. Όπως ακούσατε και στην ε, αρχή της συνεδρίασης που είχαμε την εσωτερική μας συζήτηση, ο χρόνος πιέζει και δεν θα προλάβουμε να διεκπαιρώσουμε όλα τα θέματα. Μία πολύ πολύ σύντομη, μονόλεπτη σχεδόν διακοπή για να περάσουμε στις συνέχειες ψηφοφορίες. Παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε για να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημέρης διάταξης. Την ψηφοφορία για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Σήμερα φτάνουμε στο πέρας της διαδικασίας. Θα θυμάστε ότι ο εισηγητής μας, ο κύριος Πάλλον Ντεκάστρο, μας παρουσίασε τις αδερές γραμμές της συμφωνίας ε, στις συνεδρίες της 7ης Ιανουαρίου και μάλιστα στο μεταξύ έλαβα από τον πρόεδρο της Ειδική Επιτροπής Γεωργίας του Συμβουλίου την επίσημη επιστολή που επιβεβαιώνει το, αν, το ότι αν εγκριθεί σε πρώτη ανάγνωση θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 294 της Συνθήκης και υπό την επιφύλαξη της διόρθωσης από τις νομικές υπηρεσίε. θα εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, το θέμα αυτό, σε τέτοια περίπτωση, αν το εγκρίνουμε, θα περάσει στην πρώτη ολομέλεια του Μαρτίου. Κύριε Δεκάστρο, θέλετε το λόγο? Όχι. Οπότε μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία της ε, προσωρινής ε, συμφωνίας για, την, ε, για τις θέμα της εμπορικές πρακτικές. Ονομαστική κλίση για την ψηφοφορία αυτή. Ε, ηλεκτρονικά φυσικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η προσωρινή απόφαση και συγχαρητήρια, συγχαρητήρια και πάλι συγχαρητήρια και προς τον εισηγητή, προς και εισηγητές, όλους τους συνεργάτες. Γιατί για μήνες ολόκληρους ασχοληθήκαμε με αυτό το θέμα και πραγματικά αξίζεται συγχαρητήρια. Ο κύριος Δεκάστρο έχει το λόγο. Απλά θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά όλους τους συναδέλφους. Ε, τελειώνει μια σημαντική διαδικασία. Υπενθυμίζω ότι το Συμβούλιο υπερψήφισε ομόφωνα η Ειδική Επιτροπή Γεωργίας, δηλαδή στην τελευταία συνεδρίαση πριν από λίγες μέρες, ψήφισε ομόφωνα. Είναι καλή είδηση αυτή. Σημαίνει ότι ολόκληρο το Κοινοβούλιο και ευχαριστώ τη διαπραγματευτική ομάδα ότι έκανε καταπληκτική δουλειά. Ολόκληρο το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ε, και πάλι συγχαρητήρια κύριε Δεκάστρο και σε εσά και στους συνεργάτες σας. Περνάμε στο επόμενο σημείο την εφαρμογή της έκθεσης ε, για τον κανονισμό 1 του 2005 για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά. Η συγκεκριτής μας είναι ο κύριος Ντόρμαν. Ε, θα θυμάστε ότι η Επιτροπή μας ανέλαβε από τη διάσκεψη των Προέδρων την εντολή να καταρτήσει εκτελεστική έκθεση για το πολύ ευαίσθητο θέμα της μεταφοράς των ζώων προκειμένου να διερευνήσει υποτιθέμενες παραβάσεις και κακοδιαχείριση σε σχέση με την εφαρμογή του ισχύοντος κανονισμού. Έχουμε και συνδεδεμένες επιτροπές, τις Επιτροπές Περιβάλλοντος και Μεταφορών, καθώς και την Επιτροπή Αναφορών που υπέβαλε γνωμοδότηση. 431 τροπολογίες κατατέθηκαν και 30 συμβαστικές ζήτησε το λόγο ο κύριος Νταντέν πριν δώσει το λόγο στον κύριο Τόρμαν. Όπως είπατε, είναι πολύ σημαντική αυτή η έκθεση κύριε Πρόεδρε και σε ευαίσθητη και για λόγους που με ξεπερνούν ε, διαπιστώνω το βράδυ πολύ αργά μοιράστηκε ο κατάλογος ψηφοφορίας στις πολιτικές ομάδες και Μόλις λίγες ώρες πριν την έναρξη της ε, συνεδρίασης ε, λάβαμε τις συμβαστικές τροπολογίες και έχουμε και πλέον 200 τροπολογίες που πρέπει να ψηφίσουμε πλην των, των συμβαστικών. Βέβαια μπορεί να, οι συνάδελφοι να είναι πιο έξυπνοι από μένα και πιο επιμελείς α, οι μελετηροί, αλλά εγώ δεν πρόλαβα να διαβάσω όλες τις τροπολογίες και μάλιστα ε, έχει πολλές που δεν έχουν κάνει μεταφραστήρια στα αγγλικά. Γι' αυτό ζητώ την αναβολή της ψηφοφορίας επί της εκθέσεως Ντόρμαν. Ευχαριστώ, κυρία Νόιχλ. Ich möchte dagegen reden. Θα ήθελα, αγαπητοί συνάδελφοι, να πω ότι είμαι κατά. Γιατί οι προθεσμίε είναι πολύ σφιχτέ σε όλε τι επιτροπέ. και είδατε τι γίνεται με τι διαπραγματεύσει για την ΚΑΠ. το αναγνωρίζω. Είναι πραγματικά πολύ σφιχτά τα περιθώρια, αλλά εδώ συζητάμε εκθέσεις οι οποίες θα πρέπει να κλείσουν πριν το Φεβρουάριο και αν καθυστερήσουμε θα καθυστερήσουμε και πάρα πολλά άλλα θέματα. Ελπίζω λοιπόν να καταλάβετε όλοι πως όλοι αντιμετωπίζουμε τις ίδιες πιέσεις και όλοι γνωρίζαμε πως πρόκειται για ε, προτάσεις τροπολογίας ε, που θα μπορούσαν ε, να ε, τα δούμε ένα-ένα ε, χωρίς να περιμένουμε τον κατάλογο. Άρα ναι, να ψηφίσουμε σήμερα παρακαλώ. Αγνιού. Ο κύριος Είναι η πρώτη φορά σε νέα χρόνια που έχω συμφωνήσει με τον κύριο Νταντά, αλλά όπως είπε και αυτός, οι τροπολογίες έφταναν μετά την προθεσμία σε ξένη γλώσσα. Πώς είναι δυνατόν να κάνει κανείς ε, μια σωστή επιλογή. Αν λοιπόν δεν λάβουμε θέση, αυτό θα αποτελέσει προηγούμενο, υπάρχει προθεσμία, θα έπρεπε ε, να ε, το σεβαστούμε και θα πρέπει να αναβάλουμε την ψηφοφορία μέχρι να καταφέρουμε να δούμε αυτές τις νέες τροπολογίες. Κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε σήμερα. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι βρίσκεται μέσα αυτές τις τροπολογίες. Δεν ξέρουμε τι υπάρχει στον κατάλογο ψηφοφοριών. Εάν λοιπόν ε, είναι έτσι η κατάσταση να καθυστερήσουμε, να βάλουμε την ψηφοφορία γιατί είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το θέμα. Κύριε Μαγκίνες, ευχαριστώ. Και εγώ είμαι υπέρ της αναβολής. Για τα επιχειρήματα που ακούσαμε, σημαντική πολύ έκθεση για την ε, καλή μεταχείριση των ζώων. Αλλά να μην ξεχνάμε και την ε, ευημερία των γεωργών, όχι μόνο την ευζοία, γιατί κατάγομαι από νησιωτική χώρα, είναι σημαντική η έξοδος μας προς τις αγορές και ακριβώς ε, έχω μικρό αριθμό μεγάλων μεταπίτων που θα ελέγξουν την τιμή του βοήου. Προσοχή λοιπόν. Θέλουμε υψηλέ προδιαγραφέ ε, καλή μεταχείριση και ευζοία, αλλά φοβάμαι ότι το μήνυμα αυτή τη έκθεση θα ενισχύσει του φόβου και την αβεβαιότητα των ακτινοτρόφων που εκπροσωπώ εγώ για την ε, μελλοντική κοινοτική νομοθεσία, την ώρα που το Brexit ήδη του έχει φοβήσει πολύ και η κερδοφορία ε, και τα κτηνοτροφικά και τα εισοδήματά του από την κτηνοτροφία είναι ήδη πολύ χαμηλά. Γι' αυτό είμαι υπέρ τη αναβολή. Το λόγο έχει τώρα ο εισηγητή μα, ο κύριο Ντόρμαν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα αυτό. Σίγουρα θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερο χρόνο για να ασχοληθούμε με το ζήτημα, αλλά ο Πρόεδρο αποφάσισε τα μη νομοθετικά ζητήματα, οι μη νομοθετικέ ε, εκθέσει να τι δούμε το Φεβρουάριο στο Στρασβούργο. Αλλιώ υπάρχει κίνδυνο να μην πάμε στην Ολομέλεια, αν γίνει αυτή η ψηφοφορία. Αυτή η συμβουλή λοιπόν του να ψηφίσουμε να μην υπάρξει αναβολή. Δυστυχώ δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διαθέσή μα για να ασχοληθούμε με το ζήτημα. Αλλά ήθελα να πω και κάτι άλλο. Όποιο εργάστηκε επί του θέματο αυτού είχε λάβει εν ευθέτω χρόνο έγκαιρα τι προτάσει. Είχαμε πολλού βοηθού που ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα για να κερδίσουμε χρόνο. Οι ευρωβουλευτέ που ασχολήθηκαν αν είχαν εμφανιστεί νωρίτερα, ίσως να είχαμε μπορέσει να αντιμετωπίσουμε νωρίτερα το ζήτημα. Αλλά εγώ θα έλεγα να μην ε, τα, γίνει αναβολή. Ο κύριος Ντές. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ πήρα εδώ το λόγο γιατί έχω μιλήσει με την νομική υπηρεσία και είπαμε αν αναβληθεί μέχρι την επόμενη εβδομάδα μπορούμε να το πάμε στην Ολομέλεια. Και θα ήθελα αυτός ο φάκελος να κλείσει, αλλά σήμερα δεν βλέπω πώς μπορούμε να ψηφίσουμε. Εγώ τουλάχιστον. Εγώ δεν είχα το χρόνο να εξετάσω τις προτάσεις, τις συμβιβαστικές. Λυπάμαι πολύ. Δεν έχουμε πλειοψηφία αν ε, ψηφίσουμε σήμερα, γιατί εγώ σήμερα εδώ δεν ψηφίζω. Ο κύριος Καπούτο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι πρέπει να ψηφίσουμε οπωσδήποτε ώστε να μπορέσουμε να πάμε στην Ολομελία του Φεβρουαρίου. Θεωρώ ωστόσο ότι οι παρατηρήσει των συναδέλφων ε, πρέπει να γίνουν σεβαστέ. Έχουμε περιθώριο να ψηφίσουμε και αύριο. Ίσως αυτό να είναι μια καλή ευκαιρία ώστε οι συνάδελφοι που δεν έχουν προλάβει να καθίσουν να διαβάσουν, ε, να μελετήσουν τις τροπολογίες και να ψηφίσουν αύριο. Ο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντω, ακόμη και εμεί που είμαστε μικρή ομάδα, καταφέραμε να ανταπεξέλθουμε στο φόρτο εργασία. Δεν ήταν καν φόρτο εργασία, ήταν κάπω σύντομο το χρονοδιάγραμμα. Αλλά καταφέραμε παρόλα αυτά και εξετάσαμε τι τροπολογίε. Φαντάστηκα ότι το έργο θα είχε αρκετού υπαλλήλου ώστε να μπορέσουν να, να αντιμετωπίσουν την, το έργο αυτό. Και πάνω από 200 ευρωβουλευτέ ζήτησαν τη σύσταση διερευνητική επίτροπή για το θέμα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό, θα πρέπει να το διεκπαιρεώσουμε. Και τώρα έχουμε απόφαση τη Προεδρίας για μια έκθεση εκτελεστική και αφιερώσαμε πολύ χρόνο και πολύ κόπο για την έκθεση αυτή. Και οι εκπρόσωποι του ΕΛΚΑ κατάθεσαν πάρα πολλέ τροπολογίε και προσπάθησαν να συμπεριλάβουν δικέ του ε, θέσει στην έκθεση και νομίζω ότι ήμασταν αρκετά διαλλακτικοί. Θα πρέπει να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Πάντως, αν καταφέρουμε και συμφωνήσουμε την πρόταση του κυρίου Καπούτο και αν αυτό το συμβασμό το δεχτεί το ΕΛΚ, να ψηφίσουμε αύριο δηλαδή αντί για σήμερα, δεν έχω αντίρρηση. κυρία Χάζεκαμπ. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ πολύ με τον συνάδελφο Βάιτ. Διαπραγματευτήκαμε εκτενώς και με το ΕΛΚ. Άκουσα να λένε οι συνάδελφοι και από το ΕΛΚ που ουσιαστικά γνωρίζουν λιγότερο το περιεχόμενο των συμβαστικών, παρόλα αυτά ήταν έτοιμοι. Πρέπει να πω ότι τα όσα μου είπε η κυρία Μαγκινέση μου άνοιξαν τα μάτια να διατηρήσουμε το περιεχόμενο και να σκεφτούμε και τις συνέπειες της έκθεσης. Αυτό δεν, δεν είναι λόγος για να αναβάλουμε, λέω να ψηφίσουμε. Κύριος Νίκολσον. Κύριε Πρόεδρε, όπως υπόθηκε, είναι μια σημαντική έκθεση αυτή και λεπτό θέμα, το γνωρίζουμε όλοι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα αν το αναβάλουμε για αύριο το πρωί. Αύριο 10 η ώρα. Αν μπορούμε να το συμφωνήσουμε αυτό εντό τη Επιτροπή, δεν αποτελεί πρόβλημα για μένα και ίσω τότε το ΕΛΚ να μπορέσει να δει τα πράγματα. Αλλιώ, όπω είπε και ο κύριο Βάιτ, ναι. Αν η γραμματεία μπορεί να μου επικυρώσει ότι αν δεν ψηφίσουμε σήμερα ότι αν δεν ψηφίσουμε σήμερα και δεν πάει στην Ολομέλεια του Φεβρουαρίου δεν θα συζητηθεί στην Ολομέλεια ούτε θα ψηφιστεί. Είτε δηλαδή θα ψηφίσουμε αυτή τη βδομάδα την έκθεση αυτή αλλιώ δεν θα πάει στην Ολομέλεια. Τόσο απλά. Ίσως κάποιοι να μην το θέλουν αυτό, αλλά αυτή είναι η ουσία. Αν δεν το ψηφίσουμε αυτή τη βδομάδα, ξεχάστε το, δεν πάει στην Ολομέλεια του Φεβρουαρίου θα το ρίξουμε στον Καλθόνα Χρήστον ε, για πάντα. Ε, Κύριο Σέκ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ήθελα να σας πω το εξής. Συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπε ο κύριος Βάιτς και θα σας πω γιατί. Αυτή τη στιγμή Δεν μιλάμε για τις ζάντε ενό φορτηγού ή για κάτι αμεληταίο. Μιλάμε για μια έκθεση που θα θέσει τέλος ε, ε, δυνάτων ζώων κατά τη μεταφορά. Μιλάμε για όντα ευαίσθητα. Και δεδομένου ότι η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση κολλησιεργούν εδώ και καιρό, δεν μπορούμε πια να δεχτούμε άλλες ε, ε, καθυστερήσεις. Ε, σας εκλυπαρώ. Και το ΕΛΚ είχε αρκετούς συνεργάτες για να έχει προλάβει να μελετήσει την εκθέση αυτή και τις τροπολογίες ε, μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Είναι κρίσιμο σημασία στο ζήτημα. Θα συνεχίσουν τα ζώα να υποφέρουν ή θα, επιτέλους θα κάνουμε κάτι γι' αυτό. Οπότε σας καλώ να ψηφίσουμε σήμερα. Ο κύριος Λαζά. Όντω, νομίζω ότι είναι οργανωτικό περισσότερο το θέμα. Το ΕΛΚ ε, έχει και τα μέσα και το χρόνο. Έχει πολλού βοηθού να εξετάσει εγκαίρω το ζήτημα, εμπρόθεσμα. Εμεί ε, και άλλε μικρέ ομάδε πώ καταφέραμε και τα μελετήσαμε όλα αυτά. Όντω είναι πολύ σημαντικό το θέμα και καλό θα ήταν να ψηφίσουμε τώρα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χέιτεμα. Εγώ είμαι πολύ ρεαλιστής και ζητώ να μας πει η γραμματεία ε, τι συμβαίνει και αν ε, συμφωνεί με το ότι χρειάζεται σήμερα, να, αυτή τη βδομάδα να ψηφίσουμε για να περάσουμε από ολομέλεια και αν ναι, γιατί να μην ψηφίσουμε σήμερα, γιατί να περιμένουμε μέχρι αύριο. Θα έχουμε πολλά, ε, πολύ χρόνο στη διάθεσή μας μέχρι αύριο, 12 ώρες μένουνε. Δεν μπορώ να ψηφίσω. Και επίσης χρειάζεται να φύγω. Ευχαριστώ για τα διαδικαστικά που ρώτησε η κυρία Νόιχλ και ο κύριος Βάιτς αλλά και άλλοι ευρωβουλευτές για το αν είμαστε υποχρεωμένοι να ψηφίσουμε αυτήν την εβδομάδα για να προλάβουμε να διαβιβάσουμε το ζήτημα στην Ολομέλεια του Φεβρουαρίου. Υπάρχουν κάποια όρια που μας θέτει η διάσκεψη των Προέδρων. Και γι' αυτό θα παραπέμψω το διαδικαστικό ζήτημα στη γραμματεία για να απαντήσει. Παρακαλώ, γραμματέας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω το εξής. Όντως, όπως επισήμαναν μερικοί, υπάρχει εντολή της διάσκεψης των Προέδρων ε, που μέσω επιστολής του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έλαβαν τον Ιούνιο όλες οι κοινοβουλευτικές επιτροπές και όσες ε, ακόμη έχουν εκθέσει εκθέσεις ε, ε, στο πρόγραμμά τους θα πρέπει να φροντίσουν μέχρι, μέχρι το Φεβρουάριο το αργότερο να υποβάλουν τις εκθέσεις τους για την Ολομέλεια. Οπότε αν δεν ψηφίσουμε αυτή την εβδομάδα, γιατί δεν προλαβαίνουμε την άλλη τρίτη, θα είμαστε εκπρόθεσμοι. Αν δεν ψηφίσουμε λοιπόν αυτήν την εβδομάδα, θα προλάβουμε να δώσουμε την έκθεση για την Ολομέλεια του Φεβρουαρίου. Και αν δεν προλάβουμε το Φεβρουάριο, ουσιαστικά θα είμαστε στα χέρια της διάσκεψης των Προέδρων, γιατί δεν έχουμε σεβαστεί την εντολή, τις οδηγίες, οπότε θα πρέπει να ζητήσουμε παρέκκληση και επαφή στη διακριτική ευχαίρεια τη διάσκεψη των Προέδρων, αν θα μας τη δώσει. Πάντως, επανειλημμένος, το μήνυμα και η οδηγία της διάσκεψης των Προέδρων είναι να φροντίσουμε τουλάχιστον εκθέσει πρωτοβουλία να τι διεκπαιρεώσουμε μέχρι το Φεβρουάριο, γιατί θα δοθεί προτεραιότητα για τη συνέχεια στι νομοθετικέ εκθέσει. Οπότε είναι κάπω ε, λεπτό το θέμα, αν χάσουμε αυτή την εβδομάδα. Δεύτερο, σε ό,τι αφορά την πιθανότητα να ψηφίσουμε αύριο αντί για σήμερα, αυτό γίνεται. Εσεί θα το αποφασίσετε. Αύριο το πρωί όμω έχουμε ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο Χόγκαν 9 με 10 και μισή περίπου. Γιατί λιγότερο από μια μισή ώρα αποκλείεται να φτάσει. Οπότε θα πρέπει να ψηφίσουμε αργότερα, 10 και μισή, 11 ίσως. Κάτι που προϋποθέτει τροποποίηση των υπόλοιπων σημείων της ημερήσιας διάταξης ή διεθέτηση της σειράς. Πάντως γίνεται να ψηφίσουμε αύριο αντί για σήμερα. Vamos eh, Για να δούμε λοιπόν. Εγώ δεν συμφωνώ να αναβάλουμε μέχρι αύριο. Ή θα αναβάλουμε κανονικά ή όχι αύριο. Είναι κλειστή η μερίσια ειναι κλειστη η ημερησια διαταξη και πρέπει να σας πω πως εγώ θέλω να μιλήσουμε για τις εμπορικές συμφωνίες και τις επιπτώσεις που έχουν στη γεωργία. Οπότε, με τέτοιο κατάλογο στην ημερήσια διάταξη, ε, και να χάσουμε μια ώρα με τις ψηφοφορίες από την αυριανή συζήτηση. Ή θα ψηφίσουμε τώρα ή θα το αναβάλουμε για αργότερα, όχι για αύριο. Η πρόταση για αύριο ουσιαστικά καταστρέφει τις αυριανές συζητήσεις που είναι σημαντικές. Οπότε, θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε κάτι χαλώντας τα υπόλοιπα. Οπότε, παρακαλώ, το αύριο μην το σκέφτεστε καν. Και αν δεν μπορούμε να ψηφίσουμε, ε, την επόμενη εβδομάδα ή κάποια άλλη στιγμή. Αν μπορούμε θα ψηφίσουμε σήμερα, αλλά το αυριανό δεν γίνεται, γιατί μειώνει υπερβολικά το χρόνο τη αυριανή συζήτηση. Ο κύριος Νταντάν και πάλι, ο κύριος Χόισλινγκ και τέλος. Κύριε Πρόεδρε, ακούστηκαν κάποια απαράδεκτα σχόλια. Ο καθένας δουλεύει όπως ε, κρίνει σωστό. Πρόκειται για μια έκθεση που έχει ευαίσθητο χαρακτήρα. Και δεν θα ήθελα να χωρίσω κανένα την απόφαση που πρέπει να λάβω εγώ. Δεν μπορώ α, λίγες ώρες πριν να έχω μετα, κιόλας και όλα κάποιες τροπολογίες. Έχω δικαίωμα να γνωρίζω στη γλώσσα μου ε, τις τροπολογίες. Και πριν το μεσημέρι ήμουν σε άλλη συνεδρίαση για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Ε, και η ευημερία των γεωργών είναι εξίσου σημαντικό μέλημα και προτεραιότητά μας, όχι μόνο καλή μεταχείριση των ζώων. Θέλω τουλάχιστον να σεβόμαστε το έργο των ευρωβουλευτών. Εγώ ανέκαθεν να ε, σεβόμουν το έργο των άλλων, θα πρέπει και οι άλλοι να σεβόνται το δικό μου έργο. Ο κύριος Χόισλινγκ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ πρέπει να σας πω πως θέλω να ψηφίσουμε σήμερα. Δεν ξέρω το ΕΛΚ μέσα στις επόμενες 12 ώρες τι θα καταφέρει να μάθει, αλλά έχω την εντύπωση πως πρόκειται για τακτική του ΕΛΚ που δεν, ε, δεν του αρέσει η έκθεση και δεν ξέρω αν θα του αρέσει καλύτερα αύριο. Οπότε σήμερα να ψηφίσουμε, αλλά το αργότερο αύριο. Αλλά αν υπάρχει πλειοψηφία, ψηφίσουμε τώρα. Ο Έχω μια σύντομη παρατήρηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να πω ότι εδώ πρόκειται για μια τακτική ε, κακόβουλη θα έλεγα και είμαι τελώς αντίθετο. Κύριος Ντεκάστρα, μου φαίνεται, Κάστρο, μου φαίνεται ότι η πλειοψηφία θέλει να ψηφίσει αύριο, τουλάχιστον να, να προλάβουμε απόψε να μελετήσουμε τις συμβαστικές ε, για να μην χάσουμε. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό αλλάζει λίγο την αυριανή σε διάταξη. Καταλαβαίνω, Κλάρα, αλλά είναι μια λύση συμβιβαστική που πιστεύω υποστηρίζεται από τους περισσότερους από εμάς. Ε, νομίζω ότι όλοι είχαν την ευκαιρία να εκφέρουν τη γνώμη τους. Εγώ ήμουν έτοιμος να βάλω για αύριο την ψηφοφορία, αλλά από τη στιγμή που είναι κάθετα αντίθετη η κυρία Αγγιλέρα, πρέπει να λάβουμε άλλη απόφαση. Ε, ε αύριο έχουμε πολύ φορτωμένο πρόγραμμα και κυρίως τη συνέπεια των εμπορικών συμφωνιών και της επιπτώσεις του στη γεωργία. Κάτι που ενδιαφέρει πολύ και μας και τους γεωργούς. Δεν θα πρέπει λοιπόν να περικόψουμε τη συζήτηση αυτή που είναι εξίσου σημαντική συμπεριλαμβάνοντας την ψηφοφορία. Και ε, παρόλο που ήμουν έτοιμος να προτείνω μια διαθέτηση για την αυριανή ημερήσια διάταξη για να περιλάβουμε αύριο την ψηφοφορία, μετά την ε, κατηγορηματική αντίθεση της κυρίας Αγγιλέρα, νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατο. Οπότε θα έλεγα να ψηφίσουμε. Είστε υπέρ της ψηφοφορίας του θέματος αυτού σήμερα ή αύριο. Δεν θα ήθελα εγώ να βγω από το ρόλο μου, αλλά υπάρχει μια συμβαστική λύση που θα μπορούσαμε να δούμε. Είναι αύριο. Στην ημερήσια διάταξη έχουμε τον κύριο Χόγκαν, τον Επίτροπο, και μετά μια παρουσίαση για το πρόβλημα των εσπεριδοειδών στο νότο της Ισπανίας, που είναι πρωτοβουλία της κυρίας Αγγιλέρα και έχουμε και τον κύριο Νοφρέα από τη Γενική Διεύθυνση Άγκρη που θα έρθει να μιλήσει για τα σπυριδοειδή και μετά ανταλλαγή απόψεων με τον Τζον Κλάρκ για τις εμπορικές συναλλαγές. Ίσως συμβισβασμός εδώ είναι να γίνει η συζήτηση με τον κύριο Χόγκαν, μετά η ψηφοφορία και μετά η παρουσίαση για τα σπυροειδή και να αναβάλουμε τον κύριο Τζον Κλάρκ να έρθει κάποια άλλη στιγμή. Και τα εισπεριδοειδή να τα διατηρήσουμε, γιατί ξέρουμε ότι έχουμε Ισπανούς επισκέπτες οι οποίοι το επιθυμούν. Και αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε αύριο το πρωί και μόνο να αναβάλουμε την ανταλλαγή απόψε με τον κύριο Τζον Κλάρκ, που δεν είναι, είναι ένα θέμα ενδιαφέρον, αλλά ε, όχι καυτά επί καιρό. Μάλιστα. Ε, εγώ ε, είχα την κρυφή επιθυμία να τα βολέψουμε όλα αύριο. Ε, βλέπω πάντως ότι συμφωνεί η κυρία Αγγιλέρα ανέβει, ο κύριος Χόισλεν και ο κύριος Καπρούτα επίσης ε, φαίνεται ότι συμφωνούν. Ή έχουν αντίρρηση. Όχι. Χόισλινγκ. Είχα ζητήσει εγώ να ψηφίσουμε για να ληφθεί μια απόφαση με πλειοψηφία. Θα μπορούσαμε να το είχαμε ρυθμίσει έτσι το πρόβλημα. Αλλά αν αύριο αναβάλουμε το θέμα για την εμπορική πολιτική. Ε, εγώ δεν συμφωνώ, είναι η Μερκοσούρ, ε, είναι επίκαιρο ζήτημα, δεν μπορούμε να το αναβάλουμε, ζητώ συγγνώμη. Εμένα μου δημιουργεί πρόβλημα αυτό. Ο κύριο Νίκολσον. Δεν νομίζω πως υπάρχει λόγος να τσακωνόμαστε μεταξύ μας για το θέμα αυτό. Όλοι καταλαβαίνουμε πόσο ε, πιεστικό είναι το θέμα και κατανοώ αυτούς που λένε ότι δεν είχαν το χρόνο να κάνουμε την ψηφοφορία ακριβώ μετά τον κύριο Χόγκαν αύριο στο σημείο 9 δηλαδή της ημερήσιας διάταξης και μετά ας πούμε και τα ευσπυριδοειδή γιατί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα που είναι επίγον και τις εμπορικές ε, συναλλαγές την επόμενη εβδομάδα. Γιατί πολλοί από εμά πρέπει να είμαστε σε πολλέ επιτροπές και δεν μπορούμε ξαφνικά να φύγουμε από τη μία επιτροπή για να πάμε στην άλλη. Γιατί έχουμε και άλλες προτεραιότητες είμαστε και αλλού. Οπότε προτείνω ότι όσοι είναι εδώ να ξέρουν ότι αύριο θα είναι γύρω στις 10.30 αύριο, μόλις θα έχει τελειώσει ο επίτροπος και εκείνη τη στιγμή να ψηφίσουμε τη συγκεκριμένη έκθεση. Αυτά προτείνω. Αν θεωρείτε ότι αυτό είναι απαραίτητο. Θα ήθελα όμω αύριο να ξεκινήσουμε σε νέα ακριβώ, χωρίς καθυστέρηση. Και μετά την ανταλλαγή απόψεων με τον ε, Επίτροπο θα κάνουμε την ψηφοφορία. Αν τηρήσουμε το χρόνο, θα καταφέρουμε να διεκπαιρεώσουμε όλα τα σημεία της ημερήσιας διάταξη. Θα μπορούσαμε ίσως και λίγο νωρίτερα από τις 9 να ξεκινήσουμε. Ίσως και 8.30. Πάντως ε, σας παρακαλώ να δεχτείτε αυτή την πρόταση. Κρίμα είναι να τσακωνόμαστε τώρα προς το τέλος της κοινοβουλευτική μας θητείας. Ο κύριος Χόισλινγκ. Μόνο εφόσον λοιπόν καλέσουμε τον κύριο στην Επιτροπή την επόμενη εβδομάδα. Θα προσπαθήσουμε να τον ακούσουμε αύριο τον κύριο Κλάρκ. Και αν δείξουμε επιθαρχία στην τήρηση του χρόνου στις ομιλίες θα τα καταφέρουμε. Ο κύριος Χέιτεμα. Ναι, συμφωνώ. Τα διάφορα. Μήπως να πω κάτι σήμερα για τα διάφορα, γιατί ίσως δεν προλάβω αύριο. Οπότε ολοκληρώνουμε αυτό το σημείο. Τα εσπεριδοειδή, διακόπτη κυρία Αγγιλέρα. Ναι πρώτα τα εσπεριδοειδή και μετά τα υπόλοιπα των εμπορικών συμφωνιών. Γιατί το θέμα των εσπεριδοειδών είναι πολύ σημαντικό. Αυτό πρώτα και μετά τα υπόλοιπα. Ναι, σίγουρα θα τα συζητήσουμε τα εσπεριδοειδή, οπωσδήποτε. Ωραία. Δεν έχουμε τίποτα άλλο για το σημείο αυτό. Ε, εξαντλήσαμε την ημερήσια διάταξη, λέει ο Α, συγγνώμη, ξέχασα το τελευταίο σημείο της ψηφοφορίας. Και μετά θα ακούσουμε τα διάφορα από τον κύριο Χαϊτέμα. Ε, πρέπει να ψηφίσουμε τη γνωμοδότηση της κυρίας Πετήρ. Θα ψηφίσουμε το σχέδιο γνωμοδότηση για την απαλλαγή. Δεν ξέρω αν θέλει το λόγο η συντάκτηρα της γνωμοδότησης. Καλύτερα να της το δώσω για να μας παρουσιάσει τις προτάσεις της. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους συναδέλφους που με τις τροπολογίες τους συνέβαλαν στη βελτίωση της γνωμοδότησης. Το 2017 είχαμε κάποια θετικά σημεία, λαμβάνοντας υπόψη το ελεκτικό συνέδριο, ε, την έκθεσή του για την γεωργική πολιτική. Ε, επισημάνθηκαν αρκετά προβλήματα. Θα πρέπει να εντοπίσουμε καλύτερα τα αίτια του ποσοστού σφαλμάτων της ε, ε, γεωργικής πολιτικής. Θα πρέπει ε, να λάβει υπόψη το ελεκτικό συνέδριο ότι μερικές φορές λόγω της υπερβολικής γραφειοκρατίας αυξάνεται το ποσοστό σφάλματος και δεν είναι εσκεμμένα σφάλματα. Για τα συστηματικά σφάλματα θα πρέπει να αλλάξει το σύστημα και σίγουρα θα πρέπει ε, να επιτρέπουμε απάτες κατά την ε, άσκηση των διατάξεων και την εφαρμογή των διατάξεων της κοινή γεωρικής πολιτικής. Αυτά και σας παρακαλώ να εγκρίνετε την γνωμοδότησή μου για την απαλλαγή. Σας ευχαριστούμε, οπότε περνάμε στην ψηφοφορία αγαπητοί συνάδελφοι. Είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Τροπολογία υπαριθμών 1. Διανατάσσεω της χειρός. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ. Τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση υπαριθμών 1. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ. Τροπολογία 5 υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ. 10. Α, εντάξει, ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 10. Άρχεται η τροπολογία. Otwieram głosowanie nad poprawką 10. Zamykam głosowanie. Τέλος Εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ. Εγκρίνεται. 12 υπέρ. Εγκρίνεται. 13 υπέρ εγκρίνεται. 14 υπέρ εγκρίνεται. 15 υπέρ εγκρίνεται. 16 υπέρ εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 17 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 18. Ποιο είναι υπέρ, εγκρίνεται. Και 19 υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 19, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Και ψηφίζουμε το σύνολο της γνωμοδότησης, όπως έχει τροποποιηθεί. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η γνωμοδότηση και συγχαρητήρια κυρία Πετήρ. Οπότε, αν δεν έχετε αντίρρηση, να ακούσουμε την πρόταση του κυρίου Χόιτεμα για τα διάφορα. Φαντάζομαι ότι πρώτα θέλει το λόγο ο κύριος Χαίτεμα. Ευχαριστώ πολύ. Eh, Έχω να αναφερθώ σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Πρόκειται στην πραγματικότητα για τις άδειες ε, ευρεσιτεχνίας για οποροκυπευτικά. Το 2015 ε, είχαμε ένα ψήφισμα για το θέμα αυτό. Μιλούσαμε για άδειες ευρεσιτεχνίας για τα μπρόκολα. Για ναι, μπρόκολα και για πιπεριές. Ναι, και εμείς είχαμε εκφραστεί κατά. Και οι υπουργοί το είχαν πει. Η Επιτροπή είχε πει ότι δεν ήταν αυτός ο στόχος της νομοθεσίας, ότι να χρησιμοποιηθεί η νομοθεσία αυτή για διεσέβρες τεχνές για τα προκυπευτικά. Υπήρξαν κάποιες πρωτοβουλίες, αλλά σε τεχνικό επίπεδο υπόθηκε ότι δεν υπήρχε δυνατότητα διόρθωσης. Υπάρχει αυτό ο κίνδυνος. Θέλαμε εμείς λοιπόν να μιλήσουμε με το Γραφείο Αδιώνευης Τεχνίας, να τους καλέσουμε εδώ στην Επιτροπή μας για να καταλάβουμε τι θα μπορέσουμε να κάνουμε ε, για να μπορέσουμε να ταχθούμε στο... Ευχαριστώ. Καταρχήν, κύριε Χαϊτεμα, το αίτημά σα διαβάστε το παρακαλώ στη γραμματεία για να το συζητήσουμε στη συνεδρία των συντονιστών και να δούμε αν μας το επιτρέπει ο χρόνο. Και στο μεταξύ ετοιμάστε και μια γραπτή ερώτηση για το θέμα αυτό στον αρμόδιο. Ε, το ένα δεν αποκλεί το άλλο. Γιατί έστω και γραπτός να λάβει την απάντηση χωρίς ανταλλαγή απόψεων είναι σημαντικό. Ο κύριος Χόισλινγκ. Έχουμε ήδη δύο ψηφίσματα τα οποία έχουν ψηφιστεί εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην προηγούμενη θητεία επίση. και κάθε φορά μας λέγανε πως η Επιτροπή επρόκειτο να λάβει υπόψη την ανησυχία αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έτσι ώστε να μην έχουμε τέτοιου είδου ευρεσιτεχνίε για τα τρόφιμα και τώρα συμβαίνει ακριβώς αυτό. Κάτι το οποίο μας είχαν υποσχεθεί πως δεν θα γίνει. Οπότε Πιστεύω πως θα έπρεπε εδώ να το βάλουμε στην ημερήσια διάταξη γιατί είναι πραγματικά ε, μία στάση και μία αντιμετώπιση που δεν μας αρμόζει. Εμείς είμαστε βέβαια, δεν είμαστε ε, αρμόδιοι για το τι κάνει το Γραφείο Ευρασιτεχνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά νομίζω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει, αν είμαστε σοβαροί, να εφαρμόσει αυτό το οποίο έχουμε πει δύο φορές. Και δεν είναι αρκετό με το να στείλουμε μια επιστολή. Ε, όντως επιβεβαιώθηκε η πρόταση του κύριου Χαϊτέμα. Ο κύριος Φερχούναν. Α, όχι, πρώτη κυρία Σράιερ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ήθελα να υποστηρίξω την πρόταση του συναδέλφου Γιάννη Χάιτεμα. Έχουμε μάλιστα ήδη εμπειρία με τις απαντήσεις της Κομισιόν. Συνήθως είναι συνοπτικές, πολύ. Η συζήτηση πρέπει να γίνει εδώ. Το αίτημα είναι σημαντικό, οπότε το υποστηρίζω. Εντάξει. Οπότε έχουμε τη διαδικασία τη συμφωνήσει. Άλλα διάφορα υπάρχουν. Ωραία, οπότε μπορώ να κηρύξω το πέρα στη συνεδρία της Επιτροπής Γεωργίας και να πω και πάλι ότι δεν υπήρχε καμία ιστεροβουλή, κανένας άλλο λόγο για την αναβολή ή ακύρωση της συνεδρία των συντονιστών. Ήταν πραγματικά κακή συγκυρία για παρεξήγηση. Σας διαβεβαιώ και σας δίνω το λόγο της τιμής μου ότι ζήτησα από τη Γραμματεία να κάνει γραπτές διαβουλεύσεις με τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων γιατί πραγματικά κάπως το διαστάθηκε και ζήτησε να υπάρχουν και γραπτές ε, ανταλλαγές απόψεων. Ευχαριστώ, κυρίως εδώ πέρα στη συνεδρίαση και αύριο, αύριο τα σπουδαία.